Ladies and gentlemen, nyt... Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Ας ξεκινήσουμε την ενδιαφέρουσα συνεδρίασή μας εδώ σήμερα το απόγευμα. Καλώς ορίσατε όλοι. Και φαντάζομαι ότι θα έρθουν και περισσότεροι σιγά σιγά όσο περνάει η ώρα στην αίθουσα. Βλέπετε, πολλοί από τους ευρωβουλευτές εξακολουθούν να προσπαθούν να βρουν προσπαθούν να αλλάξουν τα εισιτήριά τους εξαιτίας ε, του ηφαιστείου, προσπαθούν να βρουν άλλους τρόπους να γυρίσουν στις χώρες τους. Λοιπόν, θέλω να καλωσορίσω εδώ τους κύριους ομιλητές μας. Πρώτα απ' όλα έχουμε την κυρία Στέφανη Γκρίφιθ Τζόουνς, που είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, στη Νέα Υόρκη. Καλώς ήρθατε. Έχετε ευρεία γνώση του θέματος. Έχετε εξετάσει το θέμα της μεταφοράς κεφαλαίων στις αναδυόμενες οικονομίες. Έχετε ασχοληθεί με την μακροοικονομική διαχείριση μετακίνησης κεφαλαίων στη Λατινική Αμερική, στην Υποχοσαχάρια Αφρική επίσης. Και Επίσης έχετε εξετάσει και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις όσον αφορά τα hedge funds, τα χρηματοοικονομικά παράγωγα κλπ. Όλα αυτά λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικά για μας και γι' αυτό και χαιρόμαστε που σας έχουμε εδώ μαζί μας. Θέλω να υπενθυμίσω το εξής. Η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται στον κυβερνοχώρο. Καλό θα ήταν λοιπόν να μην μιλάτε πολύ γρήγορα όταν παίρνετε το λόγο. Θα ήταν καλύτερα να μιλάτε σε έναν ρυθμό ώστε να μπορούν οι διερμηνείς να σας μεταφράσουν. Βλέπετε έχουμε διερμηνία προς πολλές γλώσσες. Σας ακούμε λοιπόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου κάνατε να έρθω εδώ και να σας κάνω μια παρουσίαση σε αυτήν την τόσο σημαντική συνάντηση που έχετε. Θέλω να σας πω ότι τη δεκαετία του 30 υπήρχε μια αντίστοιχη επιτροπή σαν και τη δικιά σας, η οποία οδήγησε σε διάφορες μεταρρυθμίσεις στην Αμερική στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε λοιπόν μπροστά μας μια μεγάλη ευκαιρία για αλλαγές. Θέλω να σας μιλήσω για δύο ζητήματα ουσιαστικά. Και το κύριο είναι τι είδους οικονομικό σύστημα χρειάζεται η διεθνής οικονομία για να μπορέσει να υπάρξει ανάκαμψη. Πώς η Ευρώπη μπορεί να ηγηθεί αυτού του ρόλου. Θέλουμε έναν οικονομικό τομέα που να μην είναι όπως τα τελευταία χρόνια. Θέλουμε έναν οικονομικό τομέα που να αποτελεί όχι βάρος αλλά πλούτο, κέρδος για μας. Πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, πώς μπορούμε να απλοποιήσουμε, να αλλάξουμε κάποια πράγματα έτσι ώστε αντί να κυριαρχεί να εξυπηρετεί τον κόσμο και τα συμφέροντά του. Θέλω εδώ λοιπόν να ξεκινήσω με το μακροοικονομικό πλαίσιο της παγκόσμιας οικονομίας και να επικεντρωθώ κάπως περισσότερο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Νομίζω ότι, το ξέρετε και καλύτερα από μένα, ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους ο κόσμος απέφυγε την μεγάλη ύφεση σαν και εκείνη που είχαμε τη δεκαετία του 30 ήταν ακριβώς ότι υπάρχουν πολύ ισχυρέ προκυκλικές πολιτικές. Και σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα στην Κίνα, ισχύει αυτό, ότι υπάρχει μια μακροοικονομική ανταπόκριση η οποία εμπόδισε την ακόμα μεγαλύτερη κρίση. Έχουμε λοιπόν μία ανάκαμψη όπως το έθεσε και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με διαφορετικές όμως ταχύτητες. Τώρα θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει αυτή την κρίση αν ίσως δεν είχαμε ελευθερώσει τόσο πολύ το δημοσιονομικό τομέα. Έτσι καλλιώς αποφύγαμε την κρίση του 30. Οι κίνδυνοι παραμένουν διότι κάθε φορά που αποσύρονται τα αντισταθμιστικά μέτρα υπάρχει κίνδυνος για νέα προβλήματα, νέα ύφεση, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Σας αναρωτηθούμε όμως πρώτα απ' όλα, πολύ σύντομα, ποιοι ήταν οι λόγοι της επιτυχίας που είχαμε. Πρώτα απ' όλα η μαζική πολιτική παρέμβηση από τις αναπτυγμένες χώρες πρώτα απ' όλα, αλλά και από τις αναπτυσσόμενες. Δηλαδή υπήρξε μια κενησιακού τύπου ανταπόκριση από χώρες όπως ε, η Κίνα, αλλά και από άλλες αναδυόμενες οικονομίες, αναπτυσσόμενες χώρες, στις τάξεις 5-6% για να ανταποκριθούν στην κρίση. Στις αναπτυγμένες χώρες τώρα επίσης είχαμε βοήθεια από ε, τα κράτη Και επίσης πιστεύω κάτι το οποίο δεν το ακούμε συχνά. Τη στιγμή που προσπαθούμε να βοηθήσουμε και που τα θεσμικά όργανα ήταν αδύναμα, οι ηγέτες προσπαθώντας να σώσουν τις τράπεζες δεν επέβαλαν όρους για τις ρυθμίσεις. Για παράδειγμα φορολόγηση των ε, τραπεζών αυτών όταν ε, θα επανακτούσαν τα κέρδη τους. Όλα αυτά τώρα τα διαπραγματεύονται. Ο δεύτερος λόγος για την ανάκαμψη αυτή είναι η ύπαρξη μιας παράλληλης οικονομίας. Η δεκαετία του 30 βλέπετε δεν υπήρχε Κίνα όπως είναι σήμερα. Ενώ τώρα έχουμε ισχυρή οικονομία με υψηλούς δείκτες και ισχυρά οικονομικά συστήματα που μπόρεσαν να ε, λειτουργήσουν ως κίνητρο πάρα πολύ γρήγορα για την ανάπτυξη, για την ανάκαμψη μάλλον. Η Βραζιλία, η Κίνα, η Ινδία έχουν έναν μεγάλο ακόμα δημόσιο τραπεζικό τομέα. Άπαξ και πει το κράτος δανείστε περισσότερα, δανείζουν περισσότερα. Στην Κίνα, μάλιστα από ό,τι φαίνεται, οι τράπεζες δάνεισαν περισσότερα από όσα ήθελε το κράτος να έχουν δανείσει. Ένα ενδιαφέρον μάθημα είναι ότι οι χώρες αυτές και οι αναπτυσσόμενες που είχαν μεγάλο δημόσιο δημοσιονομικό τομέα όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Ινδία μπόρεσαν να ακολουθήσουν επεκτατικές πολιτικές πιστοτικές που αντιστάθμισε την μείωση των πιστώσεων σε διεθνές επίπεδο. Άλλες τώρα χώρες, η Χιλή για παράδειγμα, που είχε μια καλή πολιτική κυκλική νομισματική, εκεί δεν έγιναν τα πράγματα με τον ίδιο τρόπο, γιατί οι ιδιωτικέ τράπεζε ήταν ένα μικρό τμήμα και δεν μπόρεσαν οι πιστώσει να επεκταθούν αρκετά. Μπορούμε λοιπόν να συμπεράνουμε από όλα αυτά, από την ανάλυση αυτή, ότι η μαζική κινησιακή πολιτική δουλεύει. Ιδιαίτερα όταν οι χώρες έχουν ακολουθήσει πολύ σόφρονες μακροοικονομικές πολιτικές. Στην περίπτωση δηλαδή που έχουν περισσότερα μέσα επίσης όπως είναι, γίνεται με τις δημόσιες τράπεζες. Θέλω να επικεντρωθώ τώρα σε κάτι άλλο. Τι τύπου ε, οικονομικό σύστημα θέλουμε για να μπορούμε να, να προχωράμε σε ανάκαμψη. Μάλλον πρώτα απ' όλα τι δεν θέλουμε να έχουμε. Δεν θέλουμε να έχουμε ένα οικονομικό σύστημα το οποίο να περνάει καθετός από κρίσεις που μας κοστίζουν. Θέλουμε ένα οικονομικό σύστημα το οποίο άπαξ και υπάρξει επιβράδυνση ή μια κρίση η οποία οφείλεται είτε στο ίδιο το σύστημα είτε σε κάποιο άλλο οικονομικό σοκ να μπορεί να στηρίξει την ανάκαμψη αντί να, την επιδεινώ, να επιδεινώνει την κατάσταση. Και κατά ακόμα πιο σημαντικό, θέλουμε ένα σύστημα που να στηρίζει μια δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη, στηρίζοντας τις επιχειρήσεις, τις μικρομεσαίες ιδιαίτερα και τα νοικοκυριά, το κόσμο που έχει υποθήκες, με έναν βιώσιμο τρόπο όμως. Αυτό βέβαια κάνει τα πράγματα περίπλοκα, αλλά, ή ακούγεται περίπλοκα, αλλά δεν είναι στην πραγματικότητα. Γιατί είχαμε απλά οικονομικά συστήματα τα οποία λειτουργήσαν πάρα πολύ καλά. Ο Καναδάς το έχει ακόμα, για παράδειγμα, και η Ευρώπη το είχε στην μεταπολεμική περίοδο όταν είχε μεγάλη ανάπτυξη η Ευρώπη. Και ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες όλος παραδόξως το έχουν, ίσως γιατί έχουν, μάθει, έχουν πάρει πολλά μαθήματα από τις συχνές τους κρίσεις. Ποιοι είναι οι στόχοι τώρα. Πρέπει να έχουμε τρία μέσα πιστεύω στη διάθεσή μας. Πρώτον, ρύθμιση για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα οικονομικό σύστημα υπερβολικά φιλελεύθερο. Και πέρυσι, ε, συγγνώμη, χτες μάλλον, άκουσα τον πρόεδρο Ομπάμα, ο οποίος χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα και είπε ότι ένα μάθημα κλειδί από την κρίση αυτή είναι να προσανατολίζουμε τα οικονομικά μας και εντάξει δεν το έλεγε ακαδημαϊκά, δεν το έλεγε και οποιοδήποτε πρόεδρος των ΗΠΑ. Είπε ότι δεν είναι δυνατόν να δεχτούμε μια τέτοια κατάσταση όταν οι άνθρωποι περιμένουν δεν είναι δυνατόν να κόλλησουμε στον τοίχο, να στριμώξουμε το οικονομικό σύστημα. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ξαναδούμε ποιος είναι ο ρόλος των ε, κρατικών τραπεζών στην, ε, στο δανεισμό για να ανταποκρίνονται στις κρίσεις και όπου υπάρχουν κενά να τα καλύψουμε. Είτε δανείζοντας εμείς ήδη, είτε ενθαρρύνοντας τον ιδιωτικό τομέα να το κάνει. Στην Ευρώπη νομίζω ότι έχουμε χρήσιμα όργανα και στη Γερμανία και στην Ισπανία το ταμιευτήριο η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στην Ευρώπη που είναι ένα πάρα πολύ καλό μέσο που βοηθάει τι υποδομές και είναι κάτι που θαυμάζει ο υπόλοιπο κόσμο και όπου και αν πάω στον αναπτυσσόμενο κόσμο με ρωτάνε και θέλουν να το μιμηθούν. Και η Αμερικανική κυβέρνηση. Ένα άλλο μέσο είναι η καινοτομία που πρέπει να έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά καινοτομία, όχι έτσι όπως το καταλαβαίνει ο οικονομικός τομέας, δηλαδή να φτιάχνουμε περίπλοκα μέσα τα οποία τελικά δημιουργούν προβλήματα και έλλειψη ρευστότητας, ή οδηγούν στα τοξικά, αλλά να μπορούμε να δημιουργούμε, να επαναδημιουργούμε, εφόσον υπήρχε κατά το παρελθόν, κάτι απλό υπέρ της χρηματοδότησης. Εκκοινοπραξίες, δάνεια για τον δημόσιο τομέα, ώστε εξυπηρέτηση του χρέους να προχωράει πιο γρήγορα σε περίπτωση που πάνε καλά τα πράγματα και πιο χαμηλά σε περίπτωση που έχουμε κρίση. Ε, υποθήκες επίσης με τέτοιο τρόπο που να περιορίζουν ε, τα προβλήματα όταν βρισκόμαστε σε κρίση με ελαστικότητα, με ευελιξία. Και πάλι έχουμε παραδείγματα εδώ, τον Καναδά Όπως έλεγα και πριν λοιπόν όλα αυτά, συζητούσαμε γι' αυτό και νωρίτερα κυρία Πρόεδρε, ότι έχουμε την εντύπωση ότι είναι περίπλοκα, ότι είναι μαθηματικά μοντέλα που κανένας δεν καταλαβαίνει. Δεν είναι έτσι όμως. Πρέπει να έχουμε απλούς κανόνες. Αυτό βοηθάει. Οι οποίοι να ισχύουν επιμονή μου βάσεως, αλλά να επιδέχονται και αλλαγές εφόσον χρειάζεται, να έχουν και ελαστικότητα, που να εξυπηρετούν την πραγματική οικονομία. Γιατί αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα, το κύριο. Τέλος κύριε Πρόεδρε, θέλω να αναφερθώ λίγο και στην ρύθμιση. Με τον πρόεδρο Στίφη Σινοκάμπο ετοιμάσαμε ένα βιβλίο και θέλω να πω δύο λόγια από αυτού. Πρώτα απ' όλα, η ιστορία των οικονομικών μας δίδαξε και ο Ρόγο Βράιφεντ επίση έχει γράψει ένα βιβλίο γι' αυτό, ότι κάθε φορά που έχει κανεί μια περίοδο γρήγορου φιλελευθερισμού, έχουμε την τάση να καταλήγουμε σε κρίσεις. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι πρέπει να υπάρχουν ήδη κανόνες που να έχουν τα εξή χαρακτηριστικά. Πρώτον ότι πρέπει να είναι πλήρης, συνολική και να ισχύουν για όλους τους φορείς, για όλες τις αγορές, για όλες τις δραστηριότητες. Αν δεν το έχετε αυτό, τότε θα έχετε διατησία, αφαιρεσία και οι συστημικοί κίνδυνοι θα αυξάνονται με ταχύς ρυθμούς. Οι 20, η ομάδα των 20, το 20 συμφωνούν γι' αυτό. Αλλά βέβαια, όσοι είναι γνωστόν, ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Πώς θα γίνει αυτό, πώς θα τους έχουμε αυτούς τους κανόνες. Η ρύθμιση αυτή πάντως πρέπει να περιλαμβάνει όχι μόνο τις τράπεζες, αλλά και το σκιώδε σύστημα τραπεζών όπως το ονομάζουμε. Με ισολογισμούς που θα περιλαμβάνουμε επίσης και τα hedge funds και τις επενδυτικές τράπεζες. Τώρα εδώ η Ευρώπη και το κοινοβούλιο αυτό έχουν ηγετικό ρόλο προσπαθώντας να ρυθμίσουν τα, τις τράπεζες. Τώρα βέβαια έχουμε επιβραδυθεί λίγο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, η αλήθεια είναι ότι έχουν προχωρήσει πολύ με τα χρηματοπαράγωγα. Προσπαθούν να όμως και εκεί να τα κάνουμε περισσότερο διαφανή, ώστε να μπορούμε καλύτερα να τα ελέγξουμε. Για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα θα ήταν καλό να κάνει το ίδιο και η Ευρώπη. Η ρύθμιση πάντως πρέπει να είναι αντικυκλική. Η φιλοσοφία είναι σαφής. Και νομίζω το δεχόμαστε στην Ευρώπη αυτό περισσότερο από ό,τι στις Ηνωμένε Πολιτείες. Άρα έρχεται πρώτη Ευρώπη. Και το πρόβλημα με τις οικονομικές αγορές είναι ακριβώς το μοντέλο που ακολουθούν με μεγάλη άνοδο και ύφεση αμέσως μετά. Πρέπει να προσπαθούμε λοιπόν έγκαιρα να σταματάμε την, τον υπερβολικό δανεισμό όταν ξεπερνάει κάποια ώρα και να φροντίζουμε να υπάρχει όταν γίνεται. Όλα αυτά βέβαια μπορούν να γίνουν με κανόνες εξάντε, με των προτέρων, δηλαδή να υπάρχει από πριν η ρύθμιση. Αν δηλαδή επεκταθούν οι πιστώσει σε έναν ε, τέτοιο βαθμό, τότε κάτι κάνουμε. Και αυτός ο κανόνας να μην αλλάζει εκτός αν είναι υπερβολική επέκταση. Αν δεν το κάνετε αυτό, τότε στη μέση της οικονομικής άνθησης, και το είδαμε αυτό, με κάθε τέτοια περίπτωση, έχετε μια διαδικασία όπου όλοι λένε αυτή τη φορά θα είναι διαφορετικά. Όχι, δεν χρειαζόμαστε ρύθμιση, δεν χρειαζόμαστε να σφίξουμε τα λουριά, όχι. Ε, όχι λοιπόν, πρέπει από πριν να υπάρχει ρύθμιση, έτσι ώστε ο οικονομικός τομέας στον υπερβολικό του ενθουσιασμό να μην χάνει τον μπούσουλα και ξεπερνάει τα όρια. Για να έχουμε ένα οικονομικό σύστημα λοιπόν που να λειτουργεί υπέρ της πραγματικής οικονομίας χρειαζόμαστε καλές, απλές και αποτελεσματικές ρυθμίσεις. Πρέπει να δούμε επίσης ποιος είναι ο ρόλος ε, του κράτους και να στηρίζουμε την καινοτομία η οποία οδηγεί σε μέσα τα οποία κάνουν την χρηματοδότηση περισσότερο βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία καθηγήτρια. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία μας είπατε. Κυρία Γκρίφιθ Τζόουνς. Και ήσασταν και απλοί. Και αυτό σωστό. Τώρα περνάμε στην ε, συζήτηση. Ναι. Εντάξει, με ακούτε. Ωραία. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να δώσω τον λόγο στον κύριο Τόμασμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Γκρίφιθ ζητήσατε απλούς κανόνες. Κάνατε και κάτι άλλο. Μιλήσατε τόσο απλά για τα πράγματα που μπορούμε επιτέλους να τα καταλάβουμε. Γιατί σε μια εποχή που όλοι κρύβονται πίσω από τα λόγια, εσείς είπατε τα πράγματα απλά και σας συγχαίρω. Να εκμεταλλευτώ την ανεξάρτησία σας για να σας ρωτήσω κάτι πολιτικό γιατί είστε ακριβώς ε, μια γυναίκα η οποία δεν έχετε άμεση σχέση μπορείτε να μας τα πείτε ξεκάθαρα. Μέχρι τώρα στην πολιτική μιλούσαμε με τις ε, επιχειρήσεις και μας έλεγαν ότι αφήστε μας ήσυχους. Οπότε δεν υπήρχαν επεμβάσεις, δεν υπήρχε ρύθμιση και Τώρα εσείς μας λέτε ακριβώς το αντίθετο. Πώς πρέπει να εξυπηρετεί την οικονομία ο χρηματοοικονομικός τομέας και να υπάρχει μια ρύθμιση. Μήπως, δεν θα, έπρε... Μήπως θα έπρεπε να το δούμε πιο νωρίς αυτό. Πρόσφατα δε στις ε, είπα, συναντήθηκαν τα μεγαλύτερα αφεντικά των hedge funds με τρεις στόχους. Πρώτον, να κερδοσκοπήσουν κατά της Ελλάδος. Δεύτερον, να κερδοσκοπήσουν εις βάρος του ευρώ. Τι σημαίνει αυτό, μήπως ε, μειώνεται η επιρροή τους. Όχι. Κι όμως λέτε πως η Αμερική δεν το έκανε, δεν είναι τόσο προχωρημένη όσο εμάς. Και όμως, έτσι ήρθαν ενώπιον της γερουσίας για να δώσουν εξήγηση κάτι το οποίο δεν έγινε εδώ. Επίσης, μία πρόταση είναι να καταστρέψουμε αυτές τις τεράστιες τράπεζες. δηλαδή να έχουν τις βασικές δραστηριότητες τράπεζες και όταν δραστηριοποιούνται διεθνώς να τις επιτηρούμε. Δεύτερο ερώτημα. Εάν ε, αποφασίσει π.χ. κάτι για τα hedge funds η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν ένα ευρωπαϊκό διαβατήριο για να δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη αλλά αυτό θα έχει νόημα αν πούν και οι Αμερικάνοι α, θέμε και εμείς να ελέγξουμε τα hedge funds να υπάρχει μια διαδικασία ελεγχού ή κάπου μια καταγραφή για να δραστηριοποιούνται. Εάν κάνουμε κάτι εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύετε ότι θα ακολουθήσουν οι Αμερικανοί. Δύο φορές αναφέρατε τον Ομπάμα και ορθώς. Τι θεωρείτε, ε, μπορούμε να κρίνουμε το, το μέλλον ή ήταν μόνο ωραία λόγια. Και κατόπιν μιλάμε ήδη για διεθνή τραπεζικό έλεγχο που θα έχει νόημα όταν δεν λαμβάνει χώρα στην Ευρώπη γιατί έχουμε ταμεία εδώ πέρα αλληλεγγύης των τραπεζών. Μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό. Σε κάποια κράτη-μέλη λένε τράπεζες εμείς δεν παίζαμε σε αυτή τη ρουλέτα. είναι θεωρείται αυτές οι διαδοχικές κατηγορίες ε, είναι λογικό να γίνονται δηλαδή αφενός να κατηγορούμε τις τράπεζες και αφετέρου να τις ε, σώνουμε και τι θεωρείτε πως θα κάνουν οι Αμερικανοί uh, Έχετε τον λόγο πρώτα απ' όλα να με συγχωρέσετε το αεροπλάνο μου καθυστέρησε πάνω από μία ώρα και φαίνεται από σήμερα υπάρχει χάος στις πτήσεις έχει κλείσει το αεροδρόμιο. Ήμουν τελευταίο σου μπήκα. Εν πάση περιπτώσει έχετε τον λόγο. Φυσικά σας σεβάστηκε το ηφαίστειο. Μπράβο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την ερώτηση, η οποία είναι και δύσκολη και μπαίνει στην καρδιά του προβλήματος. Σε μια τέτοια χρονική στιγμή εσείς πρέπει να παίξετε ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Να είσαστε ανεξάρτητοι, να παραμείνετε ανεξάρτητοι και να μην υποκύψετε στα συμφέροντα διαφόρων μερών. Να ακούσετε βεβαίως ε, τις απόψεις. Εγώ ας πούμε ανήκω σε μια επιτροπή που συζητάει το θέμα αυτού του διεθνούς τέλους. Όταν μιλάμε με τις τράπεζες μας λένε αδύνατον να το εφαρμόσουμε, αλλά εμείς ξέρουμε ότι μπορούμε να το εφαρμόσουμε αυτό το διεθνές τέλος. Το ίδιο συμβαίνει και με τους κανόνες, το ίδιο συμβαίνει και με οτιδήποτε θα περιστύλει την κερδοφορία βραχυπρόθεσμα. Αλλά αν θέλουμε να τα δούμε τα πράγματα έτσι βραχυπρόθεσμα, από ευρωπαϊκή σκοπιά ή από εθνική σκοπιά ή από τη σκοπιά του απλού πολίτη, νομίζω ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ένα καλά ρυθμισμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αυτό είναι προ όφελο τη εκάστοτε χώρα. Και αν η Ευρώπη θέλει να τα βγάλει πέρα και να είναι ανταγωνιστική στην παγκόσμια αγορά, χρειάζεται ένα καλά ρυθμισμένο χρηματοπιστωτικό τομέα. Και νομίζω ότι στο μέλλον ο κόσμος θα προτιμάει να επενδύει, να αποταμιεύει και θα εμπιστεύεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα μόνο αν ε, είναι καλά ρυθμισμένο. Έχετε δίκιο που λέτε ότι ο συντονισμός με τις Ηνωμένε Πολιτείε είναι σημαντικό. Σημαντικός. Αλλά είναι ένα πρόβλημα εδώ πέρα. Βρισκόμαστε σε αδιέξοδο ούτως ή άλλως στις οικονομίες. Στις Ηνωμένε Πολιτείε λέμε ότι δεν θα πρέπει να ρυθμίζουμε ε, εμεί, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν κάνουν τίποτα. Δεν ρυθμίζουν το χρηματοπιστωτικό του σύστημα. Ίσως το ίδιο λένε και Σιγκαπούρη. Ε, νομίζω ότι πρέπει να σκεφτούμε παγκόσμια και μακροπρόθεσμα. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει ε, ένα διεθνώς ρυθμισμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αλλά αυτά που υπενηχθήκατε είναι σωστά. Ε, είναι γεμάτα όραμα. Θα πρέπει να κινηθούμε το συντομότερο δυνατό. Στο μεταξύ όμως η Ευρώπη μπορεί να πάρει το προβάδισμα ρυθμίζοντας και πλαισιώντας καλύτερα το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Παραδείγματος χάρη, αν εκφράσει ανησυχίε μέσω αυτού του κοινοβουλίου ότι πρέπει ας να ρυθμίζουμε τα hedge funds από προληπτική άποψη, νομίζω ότι μπορεί να μάθει, μπορεί να διδαχθεί ε, και η χώρα των ΗΠΑ. Επίσης, ε, θα πρέπει να υπάρχουν και κεφαλαιακές απαιτήσει για τα ίδια τα ταμεία, για τα επενδυτικά ταμεία. Ε, υπάρχει ανάγκη να προωθήσουμε πρωτοβουλίες, ε, να προωθήσουμε όσο μπορούμε το συντονισμό. Αλλά να μην αφήσουμε την έλλειψη συντονισμού να μας καθυστερήσει, γιατί τότε θα οδηγηθούμε σε παράλυση. Και τότε θα το χρησιμοποιήσει αυτό το στοιχείο ο χρηματοπιστωτικό τομέα για να μα εμποδίσει να κάνουμε οτιδήποτε. Ε, θα μας πει μην κάνετε τίποτα μέχρι να συμφωνήσετε πλήρω. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι πλήρη συμφωνία δεν θα ποτέ. Επομένω, θα πρέπει να κινηθούμε βαθμιδών, σταδιακά. Το δεύτερο ερώτημά σα αφορούσε τα ταμεία αλληλεγγύη. Νομίζω ότι οι τράπεζε θα πρέπει να συνεισφέρουν μέσω ενό φόρου ή τέλου. Με κάποιο τρόπο, εν πάση περιπτώσει. Και μέσω υψηλότερων κεφαλιάκων απαιτήσεων ε, και υψηλότερων αποθεματικών για να αποφύγουμε με μελλοντικές κρίσεις. Γιατί ξέρουμε στην τελική ότι αυτές οι τράπεζες, επειδή είναι σημαντικές για το σύστημα, θα πρέπει να τις διασώσουμε όταν υπάρχει κρίση. Και ποιος θα πληρώσει, ο φορολογούμενος. Επομένως, όσο περισσότερα κεφάλαια προβλέπουμε, ε, μέσω των κεφαλαιακών απαιτήσεων, τόσο καλύτερα, τόσο πιο ε, προστατευμένοι είμαστε θα πρέπει να υπάρχουν αποθέματα που δεν μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε ούτε για τα μπόνους, ούτε για να μοιράζουμε μερίσματα. Μέχρι το κεφάλαιο να είναι στεναρό επαρκώς. Και μόνο τότε μπορούμε να μοιράζουμε μερίσματα κτλ. Και επίσης θα πρέπει να ρυθμίσουμε και τις αποδοχές, τις απολαβές. Hans Peter Martin, ο επόμενος. Ευχαριστώ πολύ κυρία καθηγήτρια. Είναι ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέτε γιατί αν κατάλαβα καλά μας λέτε πως δεν είναι τόσο πολύπλοκα τα πράγματα πρέπει απλά να ορίσουμε ξεκάθαρους ε, κανόνες είπατε πως ε, δεν πρέπει να ρυθμίσουμε μόνο γενικά και ισοδύναμα αλλά και αντικυκλικά. Να αναφερθώ στο πρώτο σημείο. Όπως ξέρετε έχουμε μια εντονότατη συζήτηση. Επενέσατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά επιμείνατε πως θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι από το σύστημα των σκιωδών τραπεζών μέχρι τις επενδυτικές τράπεζες και τα hedge funds πώς ε, από αυτά τα οποία αντιλαμβάνεστε το τι κάνουμε αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό επίπεδο κυρία καθηγήτρια θα λέγατε πως είμαστε στο σωστό δρόμο ή βλέπετε πως οι εξελίξεις που προδιαγράφονται τώρα εδώ μέσα στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν μία, ως μία υποχώρηση και ότι κινδυνεύουμε πάλι να αφήσουμε αρκετά παραφυράκια σε όλους αυτούς τους τομείς στους οποίους εσείς ε, ζητάτε μία ρύθμιση. Γνωρίζετε την έκθεση Γκοζέ, γνωρίζετε ίσως τις τροπολογίες γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της προσποτάσει νομοθεσίες και μην ε, αισθάνεστε την ανάγκη να μας ε, επενέσετε, έχουμε σοβαρά προβλήματα. Δεύτερο ερώτημα όσον αφορά τα παράγωγα, αναφέρατε πως ε, η ΕΠΑ είναι μπροστά από την Ένωση. Κατά την άποψή σας ως επιστήμον και ανεξάρτητη, τι ε, μπορούμε εμείς ε, ως Επιτροπή να λάβουμε ως πρωτοβουλίες και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση να νομοθετήσει. Δύσκολες ερωτήσεις, λέει η κυρία Καθηγήτρια. Δεν έχω μελετήσει όλη την νομοθεσία, προσπαθώ να την παρακολουθήσω. Αλλά ε, βλέπω τώρα κάποιες αντικυκλικές προτάσεις και νομίζω είναι κατά των πολύ συγκεκριμένων κανόνων και όπως είπα θεωρώ το να έχουμε κανόνες εξάντε όπως στην Ισπανία έχει μεγάλα πλεανεκτήματα και νομίζω επίσης ότι προσπαθούν να συμμορφωθούν με τους κανόνες λογιστικής κάτι το οποίο είναι περίπλοκο αλλά πρέπει πρώτα η ε, σταθερότητα να υπερισχύσει των ε, κανόνων των λογιστικών που απευθύνονται πρώτον έγιναν στο παρελθόν και δεύτερον απευθύνονται στους επενδυτές. Στον δε τομέα των hedge funds κάνετε μια καλή αρχή αλλά τώρα επιβραδύνθηκε η διαδικασία έσβησε το μικρόφωνο της κυρίας καθηγήτριας. Well, oh, maybe use this one here. Okay, sorry. Ah, okay. Exactly, exactly. I think ναι, ναι, η επιβράδυνση ήταν που λέγαμε. Πράγματι είναι ύποπτη αυτή η διακοπή. Λοιπόν, νομίζω πως ε, τα ίδια τα hedge funds είναι σημαντικά, αλλά είναι και η ανάγκη να διατηρηθεί μια ορμή, όπως είπατε κι εσείς, για να κινηθούμε προς ένα πιο συνολικό σύστημα ρύθμισης. Δηλαδή είναι σαφές στη ΣΥΠΑ πως υπήρχε ένα όριο στον λόγο μόχλευσης για τράπεζες. Και μετά το χαλάρωσαν, κάτι το οποίο δεν έκανε ο Καναδάς και τα αποτελέσματα είναι σαφή, γιατί στον Καναδά δεν έχουν προβλήματα με τις επενδυτικές τράπεζες, ενώ είχαν σοβαρά προβλήματα στη ΣΥΠΑ. Οπότε νομίζω πως υπάρχει ανάγκη να χωρίσουμε σε αυτό το μέτωπο. Όσον αφορά τα παράγωγα, οπωσδήποτε είναι περίπλοκος τομέας, πρέπει να σκεφτούμε λίγο και σβήνει ξανά το μικρόφωνο της κυρίας καθηγήτριας. This one is working Τώρα δουλεύει το άλλο. Ε, ε δύσκολο. Λοιπόν, νομίζω όσον αφορά τα παράγωγα, ως περίπλοκος τομέας, η εντύπωσή μου είναι πως κάποια παράγωγα που είναι πολύ περίπλοκα και δημιουργούν συστημικό κίνδυνο και δεν έχουν τόσο σημαντικά θετικά μικροοικονομικά αποτελέσματα, πρέπει να σκεφτούμε το εάν έχουν κοινωνική χρησιμότητα και πως θα έπρεπε να απαγορευτούν όλος διόλου. Ναι, αλλά μπορείτε να τα, τα διαχωρίσετε. Μπορείτε να διαχωρίσετε τα κοινωνικά χρήσιμα παράγωγα και να κάνετε τη διάκριση μεταξύ αυτών και των λοιπόν. Νομίζω πως γίνεται. Προφανώς είναι ε, περίπλοκο και ίσως να υπάρχει ε, κάποιο μικροοικονομικό κόστος, κάποιος αγρότης να μην μπορεί να καλυφθεί σε κάποια πολύ περίπλοκη ε, εξαγωγή. Αλλά μπορεί αυτό να γίνει μέσω τρίτων. Αλλά πράγματα τα οποία δημιουργούν προβλήματα, π.χ. τα credit default swaps, τα ασφάλιστρα δηλαδή ομολόγων που κατ' ουσίαν παριστάνουν ότι κάποιος μπορεί να εγγυηθεί τα ομόλογα, κάτι το οποίο σε περίπτωση κρίσης ποτέ δεν γίνεται. Και υπάρχει μια επιτροπή και το συζητά αυτό το θέμα στη ΣΥΠΑ ξανά. Υπάρχει μια αξιολόγηση όπως των φαρμάκων. Και κοιτάμε στα φάρμακα όφελος και παρενέργειες. Και αυτό πρέπει να γίνει για την ε, προστασία του συστήματος και των καταναλωτών. Στην δε περίπτωση των ε, παραγόγων, καλό είναι να τυποποιηθούν και αυτή τη στιγμή τυποποιηθούν να πάνε στα χρηματιστήρια. Πρώτα απ' όλα για να υπάρχει διαφάνεια. Για να, ξέρουμε, για να ξέρουν και οι άνθρωποι τι γίνεται. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν 3 εκατομμύρια και να μην ε, ξέρουμε σε τι αντιστοιχούν και πώς θα ληφθούν και αποφάσεις πολιτικής. Και αφού υπάρχει αυτή η απόφαση μπορεί κάποιος να σκεφτεί να τα ρυθμίσει π.χ. να απαιτήσει κάποια όρια όπως το αντίστοιχο π.χ. των κεφαλιακών απαιτήσεων. Και ακόμα και αν δημιουργήσει αυτό κάποιο κόστος, πρώτα απ' όλα θα αποθαρρύνει την υπερβολική τους ανάπτυξη και θα μας δώσει έτσι κάποια, κάποιο μαξιλαράκι Οπότε δεν θα έχουμε πολλές δυσκολίες σε, περίπτωση, σε καιρούς δύσκολους. Και δεν νομίζω πως η αγορά μπορεί να το κάνει μόνη της. Π.χ. θυμάμαι στην Βραζιλία, στις τράπεζες με τα παραγωγά μας, έλεγαν οι τράπεζες πείτε στην κεντρική τράπεζα να μας ρυθμίσει. Και λέει, τους είπαμε, γιατί δεν το κάνετε μόνοι σας, αφού το ξέρετε. Και λέμε, εμείς δεν μπορούμε, γιατί αν το κάνουμε εμείς και δεν το κάνει ο ανταγωνισμός, εμείς θα χάσουμε όλους τους πελάτες μας. Οπότε πρέπει να γίνονται αυτά τα πράγματα μέσω ρύθμισης. Είναι τόσο απλό. Και νομίζω οι πεφωτισμένοι άνθρωποι στον τομέα των χρηματοοικονομικών θα το δουν. Κυρία Γκρίφιθ Τζόνς, είπατε πως είναι δύσκολες οι ερωτήσεις. Τα δυσκολότερα όμως έρχονται γιατί τελειώνει ο χρόνος, κλείνει εδώ ο κατάλογος. Ε, ναι, περβάνω, περβάνω, θα μιλήσεις. Έχουμε τέσσερις συναδέλφους ακόμα, θα ήθελα οι συνάδελφοι να κάνουν ερώτηση σε ένα λεπτό και αν μπορείτε να μας δώσετε μια απάντηση. Όλε Σμιτ, μετά Περβάνς, Ελίζα Φερέιρα και εγώ. Ευχαριστώ. Ε, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπατε, κύριε καθηγήτρια. Ο Ντομινίκ Στροσκόν είχε έρθει στην ε, Επιτροπή μας πριν από καμιά δυο εβδομάδες και είπε εν είδη συμβουλής ότι δεν θα πρέπει να εστιάσουμε τόσο πολύ στους κανόνες, στο regulation, αλλά στην εποπτεία. Γιατί οι κανόνες και οι ρυθμίσεις μπορούν να επιλύσουν τα προβλήματα τώρα. Ξέρουμε τα προϊόντα, υπάρχει αυστηρή νομοθεσία, αλλά στην πραγματικότητα είμαστε πίσω μονίμως από ένα κινούμενο στόχο. Μονίμως νέα προϊόντα, και εμείς οι νομοθέτες, γιατί είμαι νομοθέτης εδώ και 10 χρόνια, βλέπουμε ότι οι στόχοι αλλάζουν, είναι κινούμενοι και εμείς προσπαθούμε να τους υλοποιήσουμε συνέχεια. Τρέχουμε από πίσω. Είμαστε μονίμως 2-3 χρόνια από πίσω. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική μου ερμηνεία. Έτσι. Είμαστε 27 κράτη-μέλη. 27 κυρίαρχα κράτη-μέλη. Δεν είμαστε ομοσπονδιακό σύστημα. Οι χρηματαγορές είναι διαφορετικές από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Εσείς λέτε ότι θέλετε ένα παγκόσμιο σύστημα χρηματοπιστωτικής εποπτείας. Εμείς προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα ιονί, ας πούμε, ευρωπαϊκό φορέα που να ασχολείται με αυτά. Αλλά δεν νομίζετε ότι υπάρχουν τόσα πολλά ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν πριν. Στο κείμενό σας μιλάτε για τη σημασία της αρρύθμισης. Της πλήρους Θα Χρειαζόμαστε παραπάνω ρυθμίσεις. Δεν θα πρέπει να πούμε καλύτερα πιο προσαρμοσμένους κανόνες, πιο κατάλληλους κανόνες. Μήπως αυτή είναι η λέξη κλειδί. Συμφωνώ με αυτά που είπατε για την εποπτεία. Μια άλλη αποτυχία είναι ότι και με τους κανόνες που είχαμε δεν τα καταφέραμε γιατί τους εφαρμόζαμε. Στην περίπτωση του SEC, του Μέρντοφ κτλ. Δεν εφαρμόστηκαν οι κανόνες. Απέτυχε η Επιτροπή Κελφαλαιογοράς. Ε, στην περίοδο της αυτορύθμισης του Ηνωμένο Βασίλειο, ο κόσμος δεν ήθελε καν να υπάρχουν ρυθμιστικές αρχές, δεν ήθελε να ξοδεύει ούτε ένα ούτε μία πένα για να δημιουργηθούν ρυθμιστικές αρχές. Το να υπάρχει σοβαρή εποπτεία είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Το να ξέρουμε τι συμβαίνει στις χρηματαγορές, να παρακολουθούμε εκ του σύνεκης αυτούς τους κινούμενους στόχους. Και προσπαθούμε και θα πρέπει να προσπαθούμε να επηρεάσουμε την διαδικασία καινοτομία και ενδεχομένω να σπάσουμε, να μπλοκάρουμε κάποια επιβλαβή, α πούμε, νέα προϊόντα. Τώρα για την ευρωπαϊκή ή παγκόσμια ρύθμιση. Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το απαντήσω σε 30 δευτερόλεπτα. Όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχει αυτή η τάση, γιατί έχουμε τις εθνικές κυβερνήσεις, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε ευρωπαϊκές αρμοδιότητες, ενώ από την άλλη οι θεσμοί, οι φορείς είναι παγκόσμιοι. Ας πούμε σε κάποιες χώρες έχουμε ε, συνεταιριστικές τράπεζες, στη Γερμανία ας πούμε, σε κάποια lender έχουμε τράπεζες που δανείζουν ας πούμε σε τοπικό επίπεδο. Ε, δεν θα πρέπει να επηρεάζονται από τις ε, ευρωπαϊκές ρυθμίσεις, ούτε βέβαια από, και από τις ε, παγκόσμιες. Αν έχουμε όμως ε, μεγάλες τράπεζες ή μεγάλα hedge funds ας πούμε, ε, που κάνουν παγκόσμιες συναλλαγές, Αυτέ οι αγορές εξορισμού είναι παγκόσμιες. Τότε χρειαζόμαστε είτε πολύ σοβαρό συντονισμό, γιατί οι κυβερνήσεις νομίζω μπορούν να κερδίσουν αν συντονιστούν και συνδυάσουν τις κυριαρχίες τους, τι εθνικές κυριαρχίες τους. Επομένως συμφωνώ, δεν θέλουμε περισσότερη, περισσότερες ρυθμίσεις, αλλά πιο αποτελεσματικές ρυθμίσεις, πιο ευέλικτες ρυθμίσεις. Τώρα θα ακούσουμε την Περανς Περές και την Ελίζα Φερέιρα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ για όλα όσα μας είπατε, πολύ χρήσιμα. Πώς μπορούμε να οργανώσουμε τη συζήτηση, ούτω ώστε ο στόχος που μας περιγράφεται, που πιστεύω ότι συμμεριζόμαστε όλα τα μέλη της Επιτροπής και ελπίζω και του Κοινοβουλίου. Δηλαδή, αν φτιάξουμε, ξαναφτιάσουμε χρηματαγορές, θα πρέπει να εξυπηρετεί τις ανάγκε των ανθρώπων και την πραγματική οικονομία και τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να οργανώσουμε τη συζήτηση, ούτω ώστε αυτό το θέμα να τίθεται ξανά και ξανά. Γιατί η Επιτροπή της Βασιλείας κάνει ό,τι θέλει, η Ευρώπη έχει τις απόψει της και στην Επιτροπή Βασιλείας κανένας δεν προωθεί τα επιχειρήματα ε, υπέρ των μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Εγώ συζήτησα με πολλά άτομα ε, για αυτό το θέμα. Και μου είπαν, α, ξέρετε, στο G20 τα συζητάμε αυτά τα θέματα. Ο Ομπάμα μάλιστα ε, στα πλαίσια του G20 είπε τελείως διαφορετικά πράγματα σε σχέση με αυτά που είχε πει για την αύξηση των κεφαλαιακών απαιτήσεων κτλ. Πώς μπορούμε λοιπόν εμείς να θέσουμε σωστά τη συζήτηση και σε ποιο φόρουμ, σε ποιο πλαίσιο και κάποιο άλλο θέμα που δεν θέσατε. Ε, και θα ήθελα να μου να με διαφωτίσετε, γιατί είσαστε επαΐουσα. Τι θα κάνουμε με τους φορολογικούς παραδείσους, τι θα κάνουμε, πώς θα τους αντιμετωπίσουμε, πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Αν θέλουμε αποτελεσματική ρύθμιση, γιατί τη χρειαζόμαστε, το πιστεύω αυτό ότι χρειαζόμαστε, πρέπει να ανησυχήσουμε για την φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή και επομένως τους φορολογικούς παραδείσους. Άκουσα τα όσα είπε ο συνάδελφος ο Όλης Σμιτ για το better regulation. Ε, συνήθως ταυτίζεται με το λιγότερη ρύθμιση. Η καλύτερη ρύθμιση ισοδυναμεί με λιγότερη ρύθμιση. Δεν συμφωνώ με αυτό. Δεν χρειαζόμαστε νέα νομοθεσία. Ε, δεν υπάρχουν τομείς όπου πρέπει να πάμε πιο μακριά. Ίσως. Τελευταίος προβληματισμός. Αυτό που αναφέρατε για την προστασία των επενδυτών. Ε, και τον παραλυσμό με την υπηρεσία για την ε, διατροφική ασφάλεια. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να το προσπαθήσουμε ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο όταν δημιουργούμε νέες εποπτικές αρχές. Ας πούμε, η, η αρχή που με την εποπτεία των κινητών αξιών θα μπορούσε να ασχοληθεί με την καταχώρηση του πρωτοτύπου των χρηματοπιστωτικών προϊόντων και θα πρέπει να παρακολουθεί την εξέλιξη του εν λόγω προϊόντος, τι δυνατότητες έχει, πρέπει να μπει στην αγορά, πρέπει να το βγάλουμε από την αγορά, εφόσον προκύψει πρόβλημα. Αυτά έχω να θέσω ως παρατηρήσεις, λίγες παρατηρήσεις, λίγες ερωτήσεις, περιμένω τις απαντήσεις σας. Θα μιλήσω αγγλικά. Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για το ότι μιλάτε τόσο πολύ, τόσο σαφώς. Τώρα, θα ήθελα να ακούσω τη δική σας συνεισφορά και το τι σκέφτεστε για κάποιες άλλες πτυχές. Είπατε, σωστά, πώς ο χρηματοοικονομικός τομέας πρέπει να εξυπηρετεί την πραγματική οικονομία. Πριν πίσω όμως από την κρίση είχαμε και σοβαρά προβλήματα στην πραγματική οικονομία. Μεγάλα ελλείμματα, ανισορροπίες μεταξύ ΙΠΑ και Κίνας κυρίως. Όταν μιλάμε για στρατηγικές εξόδου, τι μαθήματα μαθαίνουμε για την πτυχή αυτή που τροφοδοτούσε την κρίση. Κατόπιν επανέρχομαι στους ε, ίσους όρους του διεθνούς ανταγωνισμού. Βεβαίως ε, πριν την κρίση είχαμε κάποια θεσμικά όργανα του Bretton Woods και παίζει κάποιο ρόλο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών, αλλά δεν ευθύθηκαν καν κάποιες από τις συστάσεις της Επιτροπής της Βασιλείας. Οπότε τι συμβαίνει. Είτε η ΕΠΑ και η Ευρώπη διαμορφώνουν τους όρους του παιχνιδιού για την επόμενη φάση ή θα κινδυνεύουμε όλοι να εξαχθούν κάποια από αυτά τα προϊόντα και να καταλήξουν αν θέλετε σε κάποιες ανερχόμενες αγορές που θέλουν να παίξουν τον ρόλο που ανέφεραν χτες οι Financial Times τον ρόλο της ανερχόμενης αγοράς και στον χρηματοοικονομικό τομέα. Μήπως λοιπόν καθυστερούμε να κάνουμε αυτή τη στρατηγική προσέγγιση. Τελευταίο ερώτημα. Πώς αναλύεται την ε, εμπειρία του FDIC στις ΕΠΑ γιατί είχε παίξει νομίζω κάποιο ρόλο και τέλος για τις ε, υπηρεσίες ε, αυτές. Γιατί βλέπουμε ότι δεν γίνεται αυτό σε ευρωπαϊκή ή αμερικάνικη βάση μόνο. Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, ίσως επιλέξω λίγο σε τι θα απαντήσω για να κρύψω κάπως την άγνοιά μου. Οι ερωτήσεις της Περβάνς ήταν πάντα πολύ καλές. Νομίζω είναι σαφές το που θέλουμε να πάμε. π.χ. η Βασιλεία πρόκειται περί ρυθμιστικής αρχής και, της, ε, και του σχετικού κλάδου δηλαδή και στόχο έχει και είναι πάντα προσανατολισμένη στο χρηματοοικονομικό τομέα. Και θεωρούμε πάντα ότι ξέρουμε τις απαντήσεις. Όχι. Επίσης, μία πρόκληση στο θεσμικό επίπεδο το πώς θα αναμίξουμε αυτούς που είναι στην πραγματική οικονομία, στην διαδικασία εταιρείε που δανείζονται, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακόμα και μεγάλες, συνδικάτα, τους συνταξιούχους, γιατί όλοι αυτοί επηρεάζονται. Υπάρχει, υπήρχε μια μεγάλη μάχη για τις αναπτυσσόμενες χώρες γιατί επηρεάζονταν. Αλλά είναι οι ίδιες ρυθμιστικές αρχές. και ίσως είναι σε χειρότερη κατασία από τις ανεπτυγμένες χώρες. Οπότε... Και βεβαίως αυτό πρέπει να γίνει για να εκπροσωπήσουν τα συμφέροντα της πραγματικής οικονομίας και επειδή ο χρηματοοικονομικός τομέας βεβαίως σκέφτεται βραχυπρόθεσμα και είναι πολύ σημαντικός για να τον αφήσουμε στους τραπεζίτες. Εγώ είπα βεβαίως συνολικότερη ρύθμιση, κάτι το οποίο εξορισμού σημαίνει να επεκταθεί σε προϊόντα ή σε τομείς όπου δεν υπήρχε. Τι εννοώ, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν πάρα πολλοί κανόνες, πρέπει να έχουμε απλούς κανόνες, ίσως να απαγορεύσουμε κάποια πράγματα, αλλά ευρεία γενικά κριτήρια. αυτό το πράγμα που συζητάμε στη ΣΥΠΑ, το ότι μερικέ εταιρείε είναι πάρα πολύ μεγάλε για να αποτύχουν κτλ. Πρέπει να διευρυνθεί αυτή η συζήτηση και να δούμε τις χρήσεις. Ε, του χρηματοοικονομικού κλάδου. Επίσης, κάνετε κάποιες άλλες σοβαρές ερωτήσεις. Δεν νομίζω ότι υπάρχει φόβος ανταγωνισμού με την Ευρώπη από τις αναψώμενες αγορές για αυτά τα τοξικά προϊόντα. Ένας από τους λόγους που δεν είχαν προβλήματα αυτή τη φορά οι αναδυόμενες αγορές είναι ήταν πάρα πολύ προσεκτικές. Δεν αγόρασαν τοξικά προϊόντα, είχαν το πλεονέκτημα του ότι είχαν απλά απλούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, οπότε δεν θα ανησυχούσα ακόμα για αυτούς. Έχουμε αυτή τη στιγμή στις αναπτυσσόμενες αγορές μια φούσκα η οποία αναπτύσσεται καθώς, καθώς βλέπουν πως αναπτύσσονται πάρα πολύ και μάλιστα κάποιες τέτοιες περιοχές έχουν λιγότερο πρόβλημα με το χρέος τους πρόχνουν πάρα πολύ χρήμα και δημιουργείται το επόμενο πρόβλημα. Και εκεί πέρα νομίζω χρειάζεται μια παγκόσμια ρύθμιση έτσι ώστε εάν είναι κάπως ψηλά τα επιτόκια, η συναλλαγματική ισονημία, τι μπορεί να γίνει στο διεθνές επίπεδο για να μειωθούν αυτές οι υπερβολικές ροές. Δύσκολο ζήτημα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ε, μου κάνετε τώρα ερωτήσεις, σοβαρά ερωτήματα για τις ανισορροπίες. Σύντομα, για ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Ένα από τα ζητήματα που μας απασχολεί και συζητάμε σε αυτό το βιβλίο είναι το εάν ε, κοιτάξτε το σύστημα στη ΣΥΠΑ ε, βασίζεται στο ότι οι ΙΠΑ ε, έχουν έλλειμμα και εκδίδουν δολάρια και όλοι τα χρησιμοποιούν και έτσι αυξάνεται η παγκόσμια οικονομία. Δεν είναι σωστό αυτός ο τρόπος, ξέρουμε από την εποχή των βιβλίων του Ρόμπερτ Τρίφιν. Αλλά δεν έχει γίνει τίποτα και υπάρχει πάλι ενδιαφέρουσα συζήτηση για το εάν μακροπρόθεσμα πρέπει να πάμε σε ένα πιο διεθνές ε, νόμισμα και σε μια επέκταση του ρόλου των ειδικών ε, τραβηκτικών δικαιωμάτων του Δουνουτού. Κάτι το οποίο έκανε το Διεθνές Νομισματικό εξέδωσε 250 δισεκατομμύρια ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα στην κρίση. Είναι ένας τομέας στον οποίο κοιτάνε οι συναδελφοί στο Κολούμπια, δηλαδή να μην παίζει, είπα, αυτό το ρόλο του καταναλωτή και αυτού ο οποίος θα έχει το έλλειμμα τελευταίας καταφυγής. Το, για τον φόρο στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί φαίνεται πως το θεωρούμε κάτι το, το ιδιαίτερο ότι δεν μπορεί να φορολογούμε αυτές τις συναλλαγές όλοι οι υπόλοιποι να βλέπουν φόρο αλλά όχι αυτές τις συναλλαγές γιατί λένε αν το κάνετε θα θα το αποφύγουμε. Και πάντα αυτό είναι το, το τυποποιημένο επιχείρημα. Τώρα νομίζω υπάρχει τεχνολογία να το κάνουμε λόγω των υπολογιστών έχουμε διακανονισμούς μέσω των κεντρικών τραπεζών, μέσω συμπράξεων ε, δημοσίου με τον ιδιωτικό. Γίνονται συνεχώς οι διακανονισμοί και θα μπορούσαμε να το βελτιώσουμε έτσι ώστε οι περισσότερες συναλλαγές να περνάνε από εκεί και είναι πάρα πολύ εύκολο να εφαρμόσουμε άρα ένα σύστημα φορολογίας αυτών των συναλλαγών και ένας πολύ μικρός φόρος ε, δεν θα αλλάξει, δεν θα μειώσει τη ρευστότητα και μπορεί να γίνει νομίζω και ανανόμισμα για το ευρώ, για τη λίρα και, και το δολάριο ιδεώδες θα ήταν και το γεν. Αλλά νομίζω πως ε, είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Και θα πονούσε λίγο ίσως τους πιο, τις πιο κερδοσκοπικές πτυχές αλλά κυρίως θα δώσει έσοδα σε κυβερνήσεις που είναι σε πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και για μια της παγκόσμια διακυβέρνηση αυτού του συστήματος. Ότμαρ. Κύριε Καθηγήτρια, Ε, έχω έτσι μια περίεργη αίσθηση γιατί έχουμε μια ανάλυση που πηγαίνει προς μια κατεύθυνση. Μιλάσατε για τον Ομπάμα. Αυτά τα οποία α, ανακοινώνει σημαίνει περισσότερους παγκόσμιους κανόνες. Αυτό σημαίνει πως θα έχει πλειοψηφία στη Γερουσία. Λέτε πως η Βασιλεία δύο ε, είναι σωστή. Τη διαπραγματεύτηκε η Αμερική αλλά δεν την εφάρμοσε. Μιλάμε αυτή τη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΣΥΠΑ. Μήπως οι κοινοί κανόνες δεν δημιουργούν κοινή εποπτεία. Τι σχέση έχει η εξάρτηση από το δολάριο είπα και εκείνας για την παγκόσμια ρύθμιση. Φτάνουν οι G20 και η Επιτροπή της Βασιλείας για να κάνουν αυτό το οποίο είπατε σωστά, δηλαδή να υπάρξουν παγκόσμιοι κανόνες και θεωρείτε πραγματικά πως υπάρχει πολιτική βούληση για να εφαρμοστούν όλα αυτά. Εγώ έχω την εντύπωση πως η πολιτική βούληση πάλι εξασθενεί από τις δημόσιες ε, δηλώσεις και πόσο και αν θα μπορέσουν τελικά αυτές τις δηλώσεις να γίνουν πραγματικότητα. I think Υπάρχει μια σύγκρουση μεταξύ της ε, ρητορίας και της πραγματικότητας. Όταν διαβάζετε τις δηλώσεις του G20, ε, μοιάζει με... μοιάζουμε θέσφατα. Α, είναι πολύ ακαδημαϊκά αυτά που λέει, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ λιγότερα, λιγότερο φιλόδοξα. Και η πολιτική, εσείς οι πολιτικοί, επειδή σκέφτεστε το μακροπρόθεσμο συμφέρον, των οικονομιών σας ε, μπορεί να παίξει ένα πολύ θετικό ρόλο ή πρέπει να παίξει ένα θετικό ρόλο. Τουλάχιστον περισσότερο από όσου δουλεύουν στο χρηματοπιστωτικό τομέα οι οποίοι ενδιαφέρονται ε, για τα βραχυπρόθεσμα μπόνου. Εσεί ενδιαφέρεστε για τι εκλογέ που θα γίνουν σε κάποια χρόνια, όχι για το τι μπόνου θα πάρετε αύριο. Και επομένω έχετε την ευκαιρία να σκεφτείτε για το πού πηγαίνει η οικονομία τη Ευρώπη αλλά και των χωρών σα. Φυσικά σήμερα τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα ε, από τη δεκαετία του 30 που όλη η ιστορία ήταν η Αμερική και ό,τι συνέβαινε στην Αμερική. Αν η Ευρώπη σήμερα πάρει το προβάδισμα, νομίζω ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει τις συνθήκες για μια παγκόσμια συνένεση. Αν όχι, θα υπάρξει εκ νέου κατακαιρματισμό. Η Ευρώπη θα πάει από εδώ, οι Ηνωμένε Πολιτείε από εκεί, οι αναπτυσσόμενε χώρε από την άλλη και θα αυξηθεί το χάο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να πάρετε, να πάρετε εδώ στην Ευρώπη το προβάδισμα. Νομίζω ότι βραχυπρόθεσμα δεν θα υπάρξει ένα παγκόσμιο σύστημα εθνιστικών αρχών, αλλά θα πρέπει παρόλα αυτά να υπάρξει περισσότερος συντονισμός. Ε, γιατί αυτό σημαίνει ουσιαστικά ε, μια παγκόσμια διακυβέρνηση χωρίς να, το, χωρίς να το λέμε. Μια άλλη δυνατότητα που ακούγεται στον αναπτυσσόμενο κόσμο είναι το εξής. Ότι αν δεν υπάρξει παγκόσμια ρύθμιση ε, αισθανόμαστε αβεβαιότητα και θα κλείσουμε τα κεφάλαιά μας, θα κατακαιρματίσουμε τις αγορές. Και υπάρχει πραγματικά ο κίνδυνος να κατακαιρματιστούν οι αγορές. Ε, να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι. Αν έχουμε το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο, α, βραχυπρόθεσμα θα είμαστε ασφαλείς. Τώρα, μιλάμε για το πλαίσιο, για την οργάνωση, αλλά ποτέ για τους ανθρώπους όταν μιλάμε για το σύστημα εποπτείας. Μπορούμε να έχουμε την καλύτερη οργάνωση, το καλύτερο οργανόγραμμα, αλλά αν οι άνθρωποι που δουλεύουν σε αυτό το σύστημα δεν είναι καλά καταρτισμένοι, δεν είναι οι σωστοί άνθρωποι, ε, θα έχουμε προβλήματα. Γιατί και τώρα έχουμε τρομερές πολιτιστικές διαφορές. Ορισμένοι είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι, άλλοι προέρχονται από την αγορά. Επομένως, πέστε μου εσείς την άποψή σας. Τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούμε να το κάνουμε ώστε να ξεπεράσουμε αυτές τις διαφορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχει ένα μοιραίο χαρακτηριστικό. Δεν βλέπει έγκαιρα τις αρνητικές εξελίξεις. Περιμένει ας πούμε να συμβεί το ατύχημα όπως συνέβη στην Ελλάδα για να συνειδητοποιήσει τι γίνεται. Ή περιμένει μέχρι να συμβεί το μοιραίο και μετά προσπαθεί εκ των υστέρων να βρει μια λύση αντί να προετοιμαστεί εκ των προτέρων εξάντε. Ε, και αυτό είναι αλήθεια και για την, τον επιμερισμό των αχθών. Αν υπάρχει ε, πρόβλημα στις α, διασυνοριακές συναλλαγές, δεν υπάρχει λύση εκ των προτέρων. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να προετοιμαστούμε καλύτερα. Νομίζω ότι Έχετε δίκιο. Το θέμα των ανθρώπων είναι ζωτική σημασία. Για παράδειγμα, θέλετε να έχετε καλά πληρωμένους ανθρώπους οι οποίοι να μην προσπαθούν με πλάγιους τρόπους. Ορισμένοι είπανε ότι οι πληρωμές πρέπει να συνδέονται με τα αποτελέσματα. Αυτό όμως είναι περίπλοκο. Όπως υπάρχουν τα μπόνους που δίνονται σε όσους δουλεύουν πολύ για μια επιχείρηση, θα μπορούσε ένα μέρος του μισθού να συνδυάζεται με την οικονομική σταθερότητα. Για παράδειγμα, στην Νέα γίνεται κάτι τέτοιο. Είναι δύσκολο φυσικά να μετρηθεί. Είναι όμως πράγματα που πρέπει να τα φροντίσουν. Πρώτα απ' όλα καλή κατάρτιση, κύρος. Είναι σημαντικά θέματα και για τους ρυθμιστές και για τους επόπτες, τους επιθεωρητές. Είπατε κι εσείς ότι δεν ήταν προετοιμασμένη η Ευρώπη. Είναι καλό λοιπόν τώρα που σας δίνετε ευκαιρία να το συζητάτε το θέμα της ρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά είναι τρομερό ε, ότι μπορεί να υπήρχε ολοκλήρωση, αγορές κτλ. Και όμως δεν ήσασταν προετοιμασμένοι. Δεύτερον, ναι, πρέπει να σκεφτείτε πολύ προσεκτικά μηχανισμούς μερισμού των βαρών σε περίπτωση κρίσης. Τώρα όλοι τα βάζουν με τους άλλους, ας πούμε, Ισλανδοί, ε, λένε ναι. Καλά, εγώ πιστεύω ότι, δεν, ότι είχαν ερμηνεύσει κάπως με πολύ νερό, πολύ χαλαρά τους κανόνες. Τελευταία ερώτηση και σας υπόσχομαι. Κύριε Κίσπερκ. Ναι, θα είμαι πολύ σύντομη. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίασή σας. Θέλω να έρθω σε μία από τις πτυχές που έχετε κι εσείς στην 34η σελίδα του... στην 23η σελίδα της... Ε, του κειμένου σας. Πρόκειται για όλη αυτή την πρόταση για την χρησιμοποίηση του ισολογισμού, ιδιαίτερα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών. Είδαμε και με την Λίμαν τι έγινε που κατέρευσε αυτά τα μέσα πώς χρησιμοποιούνται σήμερα. Ίσως αυτό πρέπει να δούμε πιο πολύ. Και πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον. Ίσως περισσότερο ακόμα για να μην υπάρξει η απορρίθμιση που είδαμε πρόσφατα. Τώρα και οι τράπεζες και τα άλλα χρηματοοικονομικά ιδρύματα πρέπει να μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν ειδικά μέσα εκτός ισολογισμού. 7.000 τέτοια μέσα είχαν. Δεν θα έπρεπε όλα να μπαίνουν στον ισολογισμό προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια, αντί να περιμένουμε εμείς ιδιαίτερα μέτρα, ιδιαίτερα μέσα. Απάντηση. Ε, μπορώ να σας απαντήσω σύντομα με ένα ναι. Οι Ισπανοί τι έκαναν. Είπαν όλα όσα είναι εκτός πρέπει να ανταποκρίνονται ε, στις ίδιες προδιαγραφές. Μπορεί να κάνουν πολλές ανοησίες οι ισπανικές τράπεζες, αλλά σε αυτό ήταν εντάξει. Υπάρχουν απλές λύσεις, όπως λέτε κι εσείς. Ναι, μπορούν όλα να είναι στον ισολογισμό. Δεν υπάρχει λόγος να μην είναι. Μόνο για το αρμπιτράζ, μόνο για αυτό είναι εκτός. Δεν υπάρχει άλλος λόγος. Να σκεφτούμε λοιπόν. πρέπει τα οικονομικά στοιχεία να εμφανίζονται με τον πιο διαφανή τρόπο, με απλούς κανόνες, τίποτα εκτός ισολογισμού, κανένα ειδικό μέσο. Και μετά βέβαια εποπτεία, από πολύ κοντά, έτσι, για να μην κρύβονται αλλιώς άλλα πράγματα. Και οι ρυθμιστές να τα προλαβαίνουν, αν είναι δυνατόν όλα αυτά. Έχω παραδείγματα σε δύο χώρες όπου με σε Εμένα, ακαδημαϊκό, και πήγα. Λοιπόν, γιατί δεν πρέπει να, γιατί να μην γίνονται οι έλεγχοι από κοντά πάντα και εκθέσεις κάθε τόσο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Γκρίφιθ Τζόνς για την τόσο ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων που είχαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας διαθέσατε το χρόνο σας. Τώρα, για το πρώτο πάνελ. Δεν θα σας τους παρουσιάσω όλους λεπτομέρως, έχετε πάρει νομίζω τα βιογραφικά του σημειώματα. Θα δώσω όμως το λόγο στον κύριο Νίκολας Χάτον πρώτα και μετά στην κυρία Λουκρέλτσια Ράιχλιν. Πόσο, πόσο χρόνο έχω, 5-6 λεπτά. Λοιπόν, Τρία πράγματα θα ήθελα να αναφέρω. Πρώτα απ' όλα, σε σχέση με αυτά τα οποία έλεγε στην άλλη Α, να το, να το, βγήκε. Όχι, κάντε πίσω, λοιπόν, μην, μην σας αποσπάσω την προσοχή. Η ανάπτυξη του συστήματος ε, του χρηματοοικονομικού στην Δύση έχει πλέον φτάσει στα όρια της ανοχής, ανοχής του. Να σας δώσω κάποια νούμερα που το αποδεικνύουν. Όσον αφορά δε τη στρατηγική εξόδου, εκεί είναι που πρέπει να βρούμε την ε, λεπτή ισορροπία, δηλαδή να μειώσουμε τα δημόσια ελλείμματα, ενώ και ο ιδιωτικός τομέας έχει τεράστια χρέη, όσον αφορά τα hedge funds. Να σας δώσω κάποια νούμερα που ε, νομίζω εγώ ότι πρέπει να ρυθμίσουμε καλύτερα τα χέρια της Φαντζέλα, αλλά δεν νομίζω πω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή αυτή έχουν επιλέξει το σωστό στόχο. Ε, να σας δείξω πως οι μεγαλύτεροι παίκτες στην αγορά των ε, παραγόγων είναι η Deutsche Bank, η Societe Generale και η BNP, γαλλικές και μια γερμανική τράπεζα. Και βεβαίω εκεί πέρα το πρόβλημα του ισολογισμού είναι πολύ χειρότερο από τα hedge funds και πρέπει να δείτε τι συμβαίνει στο γερμανικό και το γαλλικό τραπεζικό σύστημα και το βρετανικό. Όσον αφορά δε την στρατηγική εξόδου, ο μόνος τρόπος νομίζω να προχωρήσουμε αυτό που είπε ο David Cameron μίλησε για ένα πρόγραμμα μεγάλης κοινωνίας εγώ θα έλεγα ένα πρόγραμμα μεγάλης καινοτομίας γιατί ο μόνος τρόπος με τον οποίο θα δημιουργήσουμε πλούτο και ανάπτυξη την επόμενη δεκαετία είναι εάν υπάρξει εάν υπάρξουν καινοτόμα οικοσυστήματα που θα αυξάνουν την ανάπτυξη του τομέα της οικονομίας, της γνώσης και βεβαίως η τράπεζα, οι τράπεζες παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό και η ιστορία των τελευταίων 50 ετών πια ήταν η αποσύνδεση των τραπεζών από τα εθνικά αυτά ε, οικοσυστήματα καινοτομία και πλέον βγάζουν λεφτά από τα λεφτά. Αυτό οπωσδήποτε ισχύει για την Deutsche Bank και για άλλε τράπεζε. Θα σα δώσω λοιπόν κάποια νούμερα Τώρα, για το πρώτο δεν ξέρω αν μπορείτε να το διαβάσετε. Είναι από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο της McKinsey σε ένα έγγραφο με τίτλο «Χρέος και απομόχλευση». Μας δείχνει εδώ πέρα με στήλες τη σύνθεση δημοσίου και ιδιωτικού χρέους στις χώρες του G20. Βλέπετε σε μία άκρη το Βασίλειο και στην άλλη τη Ρωσία πάνω-πάνω είναι το δημόσιο χρέος, τα υπόλοιπα τρία κομμάτια είναι επιχειρηματικά χρέη, στεγαστικά χρέη και ο δανεισμός των τραπεζών. Και βλέπετε η Ιαπωνία, όπου το, το χρέος του δημοσίου, του ιδιωτικού με τομέα έφτασε τρεις φορές το ΑΕΠ στη δεκαετία του 1990 έχουμε 15 έτη απομόχλευσης και το ιδιωτικό χρέος και στην Ισπανία και στην ε, Βρετανία είναι πάνω από τρεις φορές ε, του ΑΕΠ και στη δε Γερμανία επίσης είναι πάνω από δύο φορές το ΑΕΠ. Και αρχίζει να γίνεται προβληματικό. Η μόνη χώρα που είχε αργεί ανάπτυξη του ιδιωτικού χρέου στην τελευταία δεκαετία είναι η Γερμανία, κατά 3% αυξήθηκε, οποιαδήποτε άλλη χώρα είχε μεγαλύτερη αύξηση του ιδιωτικού χρέους από ό,τι του ΑΕΠ. Οπότε, είπα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Νότια Κορέα πρέπει να απομοχλεύσουν όπως και η Ιαπωνία και επειδή αποτελούν το 1 τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ θα σημάνει αυτό αύξηση του δημοσίου χρέους, οπότε θα έχουμε πάρα πολύ αργή ανάπτυξη στην έξοδο από την ύφεση. Οπότε είναι πολύ δύσκολες στρατηγικές εξόδου στον δημοσιονομικό τομέα, αλλά και στον νομισματικό τομέα. Βλέπετε εδώ πέρα το πώς αυξάνονται, αυξάνεται οι Βρετανικές τράπεζες σε σχέση με το ΑΕΠ μετά τα της Ισλανδίας και δείτε εδώ πέρα αυτό εδώ το, τη διαφάνεια. Υπάρχει μία σχέση μεταξύ του ποσοστού των στοιχείων ενεργητικού του εμπορίου και της μόχλευσης. Και αυτό το οποίο θέλω να πω είναι πως η Deutsche Bank, όπως βλέπετε, έχει το υψηλότερο τέτοιο ποσοστό και την υψηλότερη μόχλευση. Και μοιάζει πάρα πολύ με hedge fund. Το ίδιο και η UPS, Societe General, BNP. Οι Αμερικανικέ τράπεζε για τις οποίες ανησυχούμε τόσο, JP Morgan, Bank of America, Chase και Citibank, είναι στον πάτο. Εμείς στην Ευρώπη έχουμε προβλήματα μόχλευσης και εμπορίας παραγωγών. Ανησυχούν οι Αμερικάνοι, εμεί πρέπει να ανησυχούμε ακόμη περισσότερο στην Ευρώπη. Επίση να δείτε και αυτό εδώ και αφορά τι ερωτήσει περί ρύθμισης. Κοιτάξτε εδώ πέρα, γιατί αξίζει λίγη μελέτη. Αυτό το οποίο βλέπετε είναι η αντίδραση των τραπεζών στην Βασιλεία 2. Το έχουμε ήδη δει αυτό στην έρευνα της Λίμαν που ανέφερε ένας συνάδελφος, στις έρευνες της ΕΠΑ και στις τράπεζες της Ισλανδίας και προκύπτει και από τις τράπεζες από τις έρευνες μας, χωρίς τον είπα, στην Γερουσία. Βλέπετε πως μετά τη Βασιλεία 2, του πώς αξιολογούσαν δηλαδή τον κίνδυνό του οι τράπεζες, το ελαφρύ και μπλε, και καθώς ε, είχαν το δικαίωμα να ρυθμίσουν εαυτόν γιατί είχαν τόσο φοβερές μεθόδους ε, διαχείρισης, μέσα σε μια δεκαετία οι ίδιες ακριβώς δομές θεωρήθηκαν 50% ε, ασφαλέστερες, λιγότερο ε, επισφαλείς από το παρελθόν. Οπότε βλέπετε εδώ πέρα οι μεγάλες τράπεζες οι οποίες παίζουν με τις ρυθμιστικές αρχές με τρόπο πραγματικά συγκλονιστικό. Εδώ πέρα πρέπει να δώσετε νομίζω το βάρος και η κλίμακα της δημόσιας παρέμβασης που χρειάστηκε να ακολουθήσει για ρευστότητα, τραπεζικές εγγυήσεις που θα τα πει η συνάδελφος. Δηλαδή η ιδέα ότι μπορούμε να τις αποσύρουμε τόσο γρήγορα με βάση την τρομερά κακή διαχείριση που έχει γίνει στους ολογισμούς των τραπεζών την τελευταία δεκαετία και την δομή των στοιχείων ενεργητικού και τα ελάχιστα κεφάλαια που εγγυώνται το τι κάνουν είναι πραγματικά μια ιδέα γελία. Η στρατηγική εξόδου θα είναι κέρια για το δυτικό τραπεζικό σύστημα για χρόνια. Δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ακόμα για έξοδο. Κάποια άλλα πράγματα, απορρίθμιση και βλέπετε εδώ πέρα το τι έχει κάνει στην ε, απόδοση της επένδυσης και εδώ πέρα στους μέσους μισθούς μια αύξηση κατά 40% αν δείτε δε τα υψηλά κλιμάκια των επενδυτικών τραπεζών, τα χρήματα τα οποία βγάζουν είναι απίστευτα στο σύμπαν αυτό που κατοικούν. Όσο για το από πού βγαίνουν αυτά τα λεφτά, τέσσερα δεν θα επεκταθώ. Ο μόνος τρόπος λοιπόν, και αυτό θέλω να πω, για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να αναπτύξει την οικονομία της γνώσης. Εκεί πέρα θα βρεθούν θέσεις εργασίας, εκεί πέρα πρέπει να δώσουμε τομεακή έμφαση και από εκεί πέρα έχουν προκύψει και όλες οι θέσεις εργασίας. Κοιτάξτε, στην Ισπανία, σε όλα τα κράτη-μέλη, εκεί πέρα δημιουργούνται θέσεις εργασίας. Αυτό θα το περάσουμε, θα βαρεθείτε, δεν θα βαρεθείτε, αλλά είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Το γράφημα τώρα, ο πίνακα που προσπέρασα ήταν μια περιγραφή του πώς λειτουργεί ένα οικοσύστημα καινοτομία ε, με παροχή γνώσης τεχνολογικής και επιστημονικής, ε, αλληλεπίδραση με επιχειρηματίες, πειραματισμός, πώς επιλέγονται οι ιδέες, πώς κινητοποιούνται πόροι Υπάρχουν πάρα πολλοί που κατοικούν, εν θέλετε, σε αυτό το οικοσύστημα της κοινοτομίας, επιχειρηματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, ο ρόλος των πανεπιστημίων. Uh, uh, Γιατί είναι ένα απολύτως, ένα απολύτως απαραίτητο τμήμα βεβαίως του συστήματος αυτού είναι η κινητοποίηση του κεφαλαίου και αποφεύγει τις υποχρεώσεις του. Στη χώρα μου θεωρώ το σύστημα το χρηματοοικονομικό και ασχολείται είτε με τα ακίνητα είτε με αυτά τα παράγωγα και τα λοιπά μέσα τα οποία προστατεύουν το σύστημα από το συστημικό κίνδυνο το οποίο αναφέραμε. Η άποψή μου είναι πως πρέπει να επανέλθει στον πλανήτη Γη το χρηματοοικονομικό σύστημα. Δεν μιλάμε μόνο για φορολογικούς παραδείσους και hedge funds. Πρέπει να δούμε πως ε, τα περίπλοκα αυτά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα βρίσκονται κατά κύριο λόγο στα μεγάλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν μόνο τρία στην Αμερική, αν συμπεριλάβουμε βεβαίως, Τα περισσότερα είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν συμπεριλάβουμε και την Ελβετία και πρέπει να δούμε εμείς πώς θα τα επιτηρήσουμε και θα τα ρυθμίσουμε. Λοιπόν, για να τελειώσω, νομίζω πως η στήριξη που ε, λαμβάνει το, το σύστημά μας και τα επίπεδα χρέους ε, που υποτίθεται ότι στόχο είχαν να προστατεύσουν τους δανειστές έναντι του πιστοτικού κινδύνου ή κινδύνου χρωστασίου είναι τόσο, τόσο διάφορα και το ίδιο ισχύει και για το επίπεδο εμπιστοσύνη μεταξύ τραπεζών έτσι ώστε οι διατραπεζικές εγγυήσει δεν ε, υπάρχουν. Βεβαίως χρειάζεται περισσότερο κεφάλαιο αλλά να θυμάστε πως ε, οι τράπεζες είναι πάρα πολύ έξυπνες στο να παίζουν και να στείλουν τις ρυθμιστικές αρχές όπως θέλουν. Αυτό έγινε στη Βασιλεία 1, προσπαθήσαμε και στη Βασιλεία 2 με, με διαφορετικές εθνικές δικαιοδοσίες που λένε πως δεν χρειάζομαστε εμείς, το... δεν έχουμε τόσο κεφαλιακές απαιτήσει και καταλήγουμε σαν ελάχιστο κοινό παρανομαστή. Οπότε δεν είμαι ιδιαίτερα αισιόδοξο και δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο ε, για μια δυναμική υπαρχή κεφαλαίου όπως ζητάει η Στέφανη καθώς μπορούν οι τράπεζες να προσφύγουν έναντι κατά των κεντρικών τραπεζών αν τους λένε να αυξήσουν τις κεφαλιακές τους απαιτήσεις. Μπορούν να βρουν διάφορα εμπόδια. Πρέπει λοιπόν να στηθούν τελείως διαφορετικά οι τράπεζες να διαχωριστεί η λιανική και χοντρική τραπεζική και οι από τις λοιπές δραστηριότητες όπως έχει πει ο Πολ Βόλκερ στις ΗΠΑ και ελπίζω να ακούσουμε την έκκλησή του δηλαδή τι γίνεται μεταξύ του ποια είναι η σχέση μεταξύ του χρηματοοικονομικού κόσμου και της πραγματικής οικονομίας δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι να έχουμε ένα τραπεζικό σύστημα τέτοιο έχει οδηγήσει όλα μας τα κράτη-μέλη να αναλάβουν κινδύνους ε, με την ε, υπόσχεση και ρητή πολλές φορές υπόσχεση πως υπάρχει εγγύηση του κράτους. Και οι άνθρωποι αυτοί τελικά σε προσωπικό επίπεδο βγάζουν πάρα πολλά χρήματα. Οπότε αν πιστεύουμε πως ε, η οικονομία μπορεί να προχωρήσει με την καινοτομία, πρέπει να επανέλθουν τα χρηματοοικονομικά συστήματα στην δημιουργία πλούτου. Οι μακροοικονομικές προκλήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Ανησυχώ πάρα πολύ για τον νόμο αυτό της Γερμανίας για τον περιορισμό της μεσονομικής πολιτικής καθώς αυξάνεται αυτή τη στιγμή η επιρροή της μεσονομικής πολιτικής, καθώς άρχισε να είναι αναποτελεσματική στα δεκαετία του 50 και του 60, σε μία δε οικονομία της ε, γνώμης έχει περισσότερη επιρροή μια τέτοια πολιτική. Αυτό μας το λέει και ο Λιβιέ Βλανσάρα από το Διεθνές τα Ταμείο και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την πολιτική για να οδηγηθούμε σε μια στρατηγική εξόδου και να περιορίσουμε τεχνητά τα ε, επίπεδα χρέους και του ιδιωτικού χρέους είναι μεγάλο λάθος. Για να συνοψίσω λοιπόν η διαχείριση της, της απομόχλευσης των υπερχρεωμένων μελών και του κόσμου το να επιτρέψουμε στα τραπεζικά μας συστήματα να έχουν ένα επιχειρηματικό μοντέλο που δεν θα βασίζεται σε ρητές αλλά και υπονοούμενες διασώσεις από τις κεντρικές τράπεζες, η διαχείριση της ζήτησης για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δουλειές είναι απίστευτες αυτές οι προκλήσεις για τις ΙΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δεν πρόκειται να μας ξεμπλέξουν οι Ασιάτες, γιατί κατά την άποψή μου το τραπεζικό σύστημα της Κίνας είναι εξίσου ασθενές με το δικό μας και η δυνατότητά του να συνεχίσει να είναι αγοραστής τελευταίας καταφυγής, να αντικαταστήσει τις ΙΠΑ δεδομένου και του μεγέθους που είναι πολύ μικρότερο από αυτό τον είπα και της ε, εγχώριας ζήτησης καθώς η εγχώρια ζήτηση στην Κίνα μικρότερη από την Ιταλία και είναι τόσο έθραυστο άρα το σύστημα της Κίνας και σημαίνει πως η και Ευρώπη θα πρέπει να απομισθούν την ευθύνη για τη διαχείριση της παγκόσμιας οικονομίας και των όρων και που θα δημιουργήσουν τέσσερι εργασία. Ευχαριστώ. <laughs> Σας ευχαριστώ. Ε, παρασυρθήκατε και έτσι από την ορμή των επιχειρημάτων σας. Ε, ξεπέρασα τον, το χρόνο σας, αλλά δεν πειράζει. Ευχαριστώ. Τώρα θα αλλάξω εστίαση στη συζήτηση αυτή και θα εστιάσω σε πολύ συγκεκριμένα θέματα των στρατηγικών εξόδου. Κυρίως την μείωση, σταδιακή μείωση των ειδικών μέτρων νομισματικής πολιτικής των τραπεζών ανά τον κόσμο που χρειάστηκαν όμως για να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Όλοι έχουμε δει τα αριθμητικά στοιχεία της κρίσης. Ε, είναι η πιο σημαντική κρίση από τη δεκαετία του 30. Ε, είδαμε τη βιομηχανική παραγωγή στην Ευρωζώνη, που είναι τέτοιου μεγέθους που σας δείχνει ποια είναι η κατάσταση, ε, ποια ήταν η ύφεση. Ε, η ύφεση ήταν ιδιαίτερα έντονη μετά το, την τράπεζα Lehman Brothers. Ε, αφού ξεκίνησε η ύφεση υπήρξε επιτάχυνση. Και αυτό δείχνει τη σημασία του χρηματοπιστωτικού παράγοντα που πολλαπλασιάζει το αρχικό σοκ που προέρχεται από την πραγματική οικονομία. Αλλά όπως βλέπετε έχουμε τώρα κάποια άτολμη ανάκαμψη. Ανακάμπτει η οικονομία, τα τελευταία αριθμητικά στοιχεία για την Ευρωζώνη είναι αρκετά ενθαρρυντικά, επομένως ήγηκε η ώρα για να θέσουμε το ερώτημα τι ειδικά μέτρα θα αντιμετωπίσουμε. Τώρα, για τον τομέα των υπηρεσιών, έχω κάποιες, κάποια γραφήματα. Τώρα, τι πολιτικές θα προωθήσουμε ως απάντηση. Θα παραπέμψω λιγάκι στην κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σε ό,τι αφορά τις παραδοσιακές νομισματικές πολιτικές, οι παραδοσιακές νομισματικές πολιτικές ήταν η δραματική μείωση των επιτοκίων. Βλέπετε το βραχυπρόθεσμο ε, επιτόκιο ε, για την ΕΚΤ και για την Federal Reserve ε, βλέπετε διαφορετικά καθεστώτα από τράπεζα σε τράπεζα. Η πρώτη κρίση ρευστότητα εμφανίστηκε τον Αύγουστο του 2007 και βλέπετε τις διάφορες φάσεις από εκεί και πέρα και μετά. είμαστε ήδη σε φάση αλλαγής των πολιτικών. Υπήρχαν όμως ε, ακόμα πληθωριστικές πιέσεις ε, στην οικονομία. Όταν κατέρευσε η Lehman Brothers, τότε οι κεντρικές τράπεζες συντονισμένα μείωσαν με δραματικό τρόπο τα επιτόκια. Και φτάσαμε σε μηδενικό επιτόκιο ε, όταν φτάσαμε στην φάση της παγίδας της ρευστότητας, όπως λένε οι τράπεζες. Για την ΕΚΤΑ, όπως βλέπετε, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η αντίδραση ήταν λιγάκι διαφορετική. Δεν φτάσαμε στο 0%, αλλά φτάσαμε στο 1%. Ε, υπήρξαν επικρίσεις στην εποχή εκείνη. Θα ήθελα να ερμηνεύσουμε διαφορετικά όμως κατά τη αυτά τα νούμερα, για να καταλάβουμε τι σημαίνει ε, επιτόκιο 1%, τι σήμαινε τότε και τι θα σήμαινε τώρα. Το να αυξήσουμε το επιτόκιο θα πρέπει να καταλάβουμε τι είναι αυτά τα ειδικά μέτρα τα οποία δημιουργήθηκαν τότε. Από τον Αύγουστο του 2007 μέχρι τον Οκτώβριο του 2008 είχαμε διάφορα μέτρα για τη ρευστότητα. Μετά όμως την Lehman Brothers είχαμε όχι μόνο αλλαγές στα μέτρα που αφορούσαν τη ρευστότητα, αύξηση τη ορίμαση κτλ, αλλά και αύξηση των ισολογισμών των κεντρικών τραπεζών. Όπως και άλλες κεντρικές τράπεζες ανά τον κόσμο και ο ισολογισμός της ΕΚΤ αυξήθηκε. Αυξήθηκε λοιπόν, ε, αυξήθηκαν τα στοιχεία του παθητικού. Άρα υπήρξαν μέτρα δημιουργία χρήματο. Αυτά τα μέτρα Ε, που σήμαιναν ότι θα δώσουν ρευστότητα στις τράπεζες, οι κεντρικές τράπεζες. Ε, με την αυξημένη ορίμανση στις μακροπρόθεσμες πράξεις, ε, με διατάξεις ρευστότητας σε ξένα νομίσματα και με προγράμματα αγοράς καλυμμένων ομολόγων. Όλα αυτά τα μέτρα είχαν σαν αποτέλεσμα να εξομαλύνουν τις ε, χρηματαγορές. Αυτό είναι το spread μεταξύ του LIBOR και του OIS. Είναι ένας δείκτης των τάσεων στις χρηματαγορές, έτσι βραχυπρόθεσμα. Βλέπετε το πικ ε, στη Lehman Brothers και πώς υπήρξε αυτή η μείωση μετά και που εξηγεί το επίπεδο στο οποίο έχουμε φτάσει τώρα. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο σώθηκε το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Εγώ λοιπόν είμαι λιγότερο απεσιόδοξη από τους ε, προλαλήσαντες για το πώς λειτουργήσαν αυτές οι πολιτικές. Ε, αν δείτε αυτό το πολύχρωμο ισοζύγιο, ισολογισμό μάλλον, βλέπουμε τις, τα στοιχεία του παθητικού κάτω από το 0 και τα στοιχεία του ενεργητικού πάνω από το 0. Τα ειδικά μέτρα άλλαξαν τα δεδομένα και βλέπετε χάρη σε αυτό το διάγραμμα το μέγεθος του ισολογισμού. Η πτώση μετά το, τη Λίμαν δεν σήμαινε μόνο ότι άλλαξαν οι πράξεις, αλλά και πώς επεκτάθηκαν ουσιαστικά τα ισοζύγια, τα ισολογισμοί. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα για την Fed, πολύχρωμο επίσης. Βλέπουμε εδώ ε, της ε, Κεντρικής Τράπεζας Αγγλίας τι έγινε προ και μετά την Lehman Brothers. Βλέπετε τη χρονική στιγμή, πόσο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, πόσο επεκτάθηκαν οι ισολογισμοί. Οι κεντρικές τράπεζες έγιναν μεγάλη ενδιάμεση. Ουσιαστικά αντικατέστησαν ε, τις ε, ιδιωτικές χρηματαγορές. Και αυτό είναι ένα μεγάλο ιστορικό στοιχείο. Η επέκταση των στοιχείων του αρνητικού των κεντρικών τραπεζών δεν είχαν επίπτωση στον πληθωρισμό. Λόγω του κινδύνου των χρηματαγορών και την ε, συμπεριφορά του κοινού, ξέρουμε πολύ καλά ότι ο πληθωρισμός δεν εξαρτάται μόνο από την προσφορά χρήματος, αλλά και από τη συμπεριφορά του κοινού. Επίσης, η πιστοτική υποστήριξη της ΕΚΤ δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως ε, προσφορά χρήματος, αλλά και σε σχέση με το τι κάνει στα επιτόκια. Μόνο αν καταλάβουμε αυτό το στοιχείο, μπορούμε να μιλήσουμε μετά για στρατηγικές ε, εξόδου και να καταλάβουμε τις ανακοινώσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και των υπόλοιπων κεντρικών τραπεζών. Ας δούμε τα βραχυπρόθεσμα επιτόκια της ε, Ευρωζώνης. έχουμε αυτό το επιτόκιο που είναι υψηλότερο από το βασικό επιτόκιο των αγορών. Στις περιόδους έντασης ήταν πολύ υψηλότερο και μετά έχουμε και το επιτόκιο της αγοράς. Παρότι το επιτόκιο είναι στο 1%, δηλαδή είναι ε, το επιτόκιο που προωθούν οι νομισματικές πολιτικές της ε, ΕΚΤ, το πραγματικό επιτόκιο της αγοράς είναι πολύ χαμηλότερο. Αυτό είναι αποτέλεσμα των ειδικών μέτρων που προωθεί η ΕΚΤΑ. Η νομισματική πολιτική, δηλαδή, στην πραγματικότητα ε, ευνοεί πολύ περισσότερο και προσαρμόζεται πολύ περισσότερο στην κατάσταση από ό,τι φαίνεται εκ των προτέρων. Τα spreads είναι πολύ σημαντικά για τη χρηματοδότηση των Τώρα, για το phasing out. Αυτό είναι το προφίλ διαφόρων πράξεων. που πρέπει να λάβουν χώρα ε, μέχρι το 2011. Μέχρι το τέλος του 2010 θα έχουμε υπερβολική ρευστότητα. Τον Ιούλιο είχαμε την ειδική πράξη τι τις ειδικές επιχειρήσεις που, θα σταμάτησαν και μείωσαν το βαθμό της ρευστότητα, αλλά τα προφίλ που ανακοίνωσε ο Τρισέ στην πραγματικότητα σηματοδοτούν μια πολύ προσεκτική στάση. Επομένως η ρευστότητα θα μειωθεί βαθμιδών και θα κρατήσουμε το βασικό επιτόκιο σταθερό. Λοιπόν, από μακροοικονομική προοπτική θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το policy rate, αυτό το επιτόκιο είναι σταθερό. Αλλά αυτό τι σημαίνει για την πραγματική οικονομία. Τι σημαίνει για την πραγματική οικονομία ότι τα ειδικά μέτρα ρευστότητας βαθμιδών θα καταργηθούν. Καταρχάς ότι θα προχωρήσουμε βαθμιδών. Ε, θα έχουμε πλεόνασμα ρευστότητα. Και μετά το τέλος του χρόνου μπορούμε να περιμένουμε μία εξομάλυση και κάποια επίπτωση στην πραγματική οικονομία και στα δάνεια. Δηλαδή μιλάω για το 2011 και μετά. Πόσο σημαντικές είναι αυτές οι επιπτώσεις. Πιστεύω ότι θα είναι σχετικά μικρές, αλλά όχι μηδενικές. Θα υπάρξει κάποια συρρήκνωση το 2011. Εγώ καταλαβαίνω την άποψη της ΕΚΤΑ. Καταλαβαίνω την προσέγγισή της, η οποία είναι προχωρούμε βαθμιδών. Να κρατήσουμε το επιτόκιο σταθερό και τα μέτρα ρευστότητα να τα ακυρώσουμε πραγματικά σταδιακά. Γιατί τότε λοιπόν δεν θα έπρεπε η Έκτε να παραμείνει στεναρή και να, να συνεχίζει να τροφοδοτεί τις τράπεζες με ρευστότητα. Όχι είναι η απάντησή μου. Θα πρέπει να δώσουμε μια κάποια ελευθερία στην αγορά, να λειτουργήσει από μόνη της η αγορά, να απογαλακτιστεί από την υποστήριξη των κεντρικών τραπεζών. Ένα συνάδελφος είπε ότι αυτό είναι μη ρεαλιστικό. Θα πρέπει να συνεχίζουμε να τροφοδοτούμε τις τράπεζες. Γιατί υπάρχει μια αστάθεια χρηματοπιστωτική. Εγώ όμως διαφωνώ. Υπάρχουν κάποιες τάσεις στο τραπεζικό σύστημα. Βλέπουμε ότι το, η μέση εγγραφή αυξάνεται παρότι δανειζόμαστε πιο φθηνά στην αγορά. Αυτό δεν αφορά όμως καθαρά τον τραπεζικό τομέα, αφορά διάφορους α, χρηματοπιστωτικούς φορείς. η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν καταλαβαίνετε τη λογική αυτών που λέω, ε, είναι ότι προσπαθεί να ρυθμίσει την ρευστότητα μέσω του πραγματικού επιτοκίου. Αλλά αυτά που λένε στο κοινό είναι ότι Τώρα λειτουργεί η νομισματική πολιτική με τρόπο τελείω διαφορετικό από ό,τι πριν από την κρίση. Θα πρέπει να δούμε και τα δύο επιτόκια, και το ε, αγοραίο επιτόκιο επιπλέον. Βεβαίως, αν υπάρξουν πληθωριστικές τάσεις όταν αρχίζει η ανάκαμψη της πραγματικής οικονομίας, θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Αυτό είναι σημαντικό ή έχει μόνο τεχνικό χαρακτήρα. Και ναι και όχι. Θα πρέπει να δούμε την νομισματική πολιτική σε σχέση με άλλες πολιτικές. Τέλειωσε ο χρόνος μου. Ναι, τέλειωσε ο χρόνος σας. Όταν αυξηθεί το επιτόκιο, τι θα γίνει στις αγορές. Νομίζω ότι υπάρχει χρόνος μέχρι να υπάρξει σύγκληση των δύο επιτοκίων. Αυτό όμως το ερώτημα είναι συγκυριακό. Υπάρχει ένα βαθύτερο ερώτημα που πρέπει να ρωτήσουμε. Σε αυτόν τον νέο κόσμο τι θα κάνουν οι τράπεζες, οι κεντρικές τράπεζες. Καταρχάς η ΕΚΤ δεν είναι ρυθμιστική αρχή, αλλά έχει λειτουργίες μακροπροληπτικές. Και πρέπει να θέσουμε το ερώτημα τι εργαλεία έχει η ΕΚΤ για αυτές τις ε, μακροπροληπτικές λειτουργίες. κάνει ανάλυση, ε, δίνει μηνύματα προειδοποίησης. Στην πραγματικότητα όμως και σε αυτό το επίπεδο δεν έχει πολλά εργαλεία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα για την ανάλυση και την, το κρούσιμο του κόδωνα. Και δεν υπάρχει και μεγάλη εμπειρία. Στην πραγματικά, στο εσωτερικό της ΕΚΤ πρέπει να γίνει ένας προβληματισμός για το πώς θα ασχοληθούν με το ερώτημα. Δηλαδή με το ερώτημα του ότι έχουν πολύ λίγα εργαλεία στη διάθεσή τους. Και οι σχέσεις από την άλλη, ποια είναι η σχέση με τις ε, δημοσιονομικές πολιτικές. Η, η μόνη πολιτική που μπορεί να χρησιμοποιήσει στην πραγματικότητα η ΕΚΤ και που το έκανε στην περίπτωση της Ελλάδας είναι η παράταση της πολιτικής των collateral. Το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για την ε, ζώνη του ευρώ. Με αυτά ολοκληρώνω. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Ο Hans Peter Μάρτιν είναι ο πρώτος που έχει ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι που σας έχουμε εδώ, που σας προσκαλέσαμε. Ένα πράγμα θέλω να ε, σας ζητήσω. Μπορείτε να μας αφήσετε τις διαφάνειες, φωτοτυπίες αυτών που μας είπατε. Τώρα όσον αφορά τις συστάσεις σας. Είπατε ότι το οικονομικό σύστημα απαιτεί συνεχή στήριξη για μια δεκαετία και ότι τα χρέη παντού θα αυξηθούν. Και εσείς και εγώ ήμασταν πριν δημοσιογράφοι. Τι θα μας συστήνατε τώρα που εμείς εκπονούμε πολιτική. Να πείσουμε το δημόσιο ότι είναι εφικτό. Είμαι από την Αυστρία, αλλά και με την Γερμανία συνεργάστηκα πολύ στο παρελθόν. Εσείς τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Μπορείτε να επηρεάσετε την κοινή γνώμη στη Γερμανία έτσι ώστε να σας καταλάβει χωρίς να εθνικοποιήσετε τράπεζες. Για μένα αυτό είναι το συμπέρασμα μετά από αυτά που είπατε για την έλλειψη εμπιστοσύνη, για τη συμπεριφορά των ε, τραπεζών. Σας κατάλαβα καλά ή εσείς βλέπετε κάποια άλλη λύση μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού τρόπου σκέψης για την εθνικοποίηση των τραπεζών. Να ακούσουμε και την επόμενη ερώτηση, λέει ο Πρόεδρος, και μετά να απαντήσετε. Η κυρία Κέρσμα. Ναι, ναι, κάντε την ερώτησή σας. Μα νομίζω ότι είχε και άλλη ερώτηση. Για άλλον ομιλητή, έτσι δεν είναι. Ναι, ναι. Για την κυρία Ρέχλιν έχω να ρωτήσω κάτι. Λοιπόν, για να μιλήσει γερμανικά. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, με αυτή τη σοβαρή πίεση των 420 ε, δισεκατομμυρίων που θέλει τέλος Ιουνίου να ανακαλέσει. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι έτσι θα γίνουν τα πράγματα είναι μια υπόθεση αυτά από μέρους σας. Και αν υπάρξει κάποια παράταση, τι συνέπεια θα έχει αυτό για τις γενικές σας υποθέσεις όσον αφορά αυτόν τον τομέα. Ωραία, λοιπόν, απαντήστε εσεί πρώτα. Ναι. Βεβαίω, και ευχαρίστως και τι διαφάνειε και την φωτοτυπία να σα αφήσω. Κανένα πρόβλημα. Και συγγνώμη αν δεν τα είχατε ήδη όλοι από πριν. Ε, νομίζω ότι εσείς με ρωτάτε για την περίπτωση Χάμπλινγκ, έτσι δεν είναι. Δεν νομίζω ότι το γερμανικό κοινό γνωρίζει τις λεπτομέρειες για το τι γίνεται στο τραπεζικό σύστημα. Κυρίως πρόκειται για τις τρεις μεγάλες τράπεζες που γίνονται ενεργοί παίκτες στο σύστημα Νεσιόρκης Λονδίνου. Δεν ξέρω αν και άλλη τράπεζα θα μπορούσε να συμμετάσχει. Πάντως, μία από τις προκλήσεις είναι αυτά που αντιμετωπίζουμε και στην Αγγλία και στη Γαλλία και στην Ισπανία. Και εκεί έχουμε ένα αντίστοιχο φαινόμενο, ίσως λιγότερο οξύ στην Ιταλία, όπου το τραπεζικό σύστημα διεθνοποιείται και αποσυνδέεται από την καινοτομία στο εσωτερικό της χώρας. Μόνο μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να ξεφύγετε από τις φορολογικές πολιτικές. Δεν μπορείτε να τα έχετε και τα δύο. Αλλιώ την επόμενη δεκαετία θα έχουμε τεράστια προβλήματα. Γι' αυτό και μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίαση που ακούσαμε μόλις τώρα για τις δράσεις που αναλαμβάνονται, για τις εγγυήσεις. όλα αυτά είναι φοβερά μέτρα. αν αποσύρονταν γρήγορα δεδομένης της έλλειψης εμπιστοσύνη που υπάρχει στις αγορές, δεν ξέρω αν θα ήταν τα πράγματα εξίσου καλά όπω είναι και τώρα. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Εγώ μιλάω βάσει της δωδεκάμινης εμπειρίας που έχω, ξέροντας ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό κινδύνου, αλλά υπάρχουν και διευκολύνσεις βάσει συντονιστικών δράσεων που έχουν βοηθήσει. Ό,τι σενάρια για να έχουμε δει από την αγορά και από τις μελέτες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δεν νομίζω ότι μπορούμε να περιμένουμε ρεαλιστικά μια αύξηση υπερβολικής ρευστότητας, αλλά ούτε και προβλήματα ρευστότητας μεγάλα, αν και θα υπάρξουν κάποιες εντάσεις για κάποια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για παράδειγμα τις ελληνικές τράπεζες. Η ευρωπαϊκή κατάσταση πάντως σε σχέση με το Federal Reserve, η διαφορά είναι ότι ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει χωρίς μεγάλες αλλαγές στο ρυθμιστικό πλαίσιο. Είναι εύκολο να μπει κανεί και να βγει, παρόλο που υπάρχουν και διάφορα λεπτά ζητήματα πώς αποσυρώμαστε χωρίς να δημιουργηθεί μεγάλη αστάθεια. Πάντως, αν δεν πιστεύετε ότι οι τράπεζες είναι ευάλωτες, είναι αυτό που είπατε εσείς, ναι. Δεδομένων των προσδοκιών όσον αφορά την ανάκαμψη της ε, πραγματικής οικονομίας και δεδομένης της κατάστασης της περισσότερες ευρωπαϊκές τράπεζες, νομίζω πως όχι. Και μένουμε τώρα. Ναι. Έχω και εγώ δύο διαφορετικά είδη ερωτήσεων γιατί δύο μιλητές έθιξαν διαφορετικά ζητήματα. Τους ευχαριστώ και τους δύο. Κύριε Χάτον, λέτε ότι πρέπει να έχουμε ένα καλό παράδειγμα και να υπάρχει ευθυγράμμιση ώστε να προχωρήσουμε σε καινοτομίες στο οικονομικό σύστημα. Μέχρι τώρα αυτό γινόταν από μη τράπεζες, από ε, hedge funds, από κοινοπραξίες. Πώς τώρα θα προχωρήσουμε ενθαρρύνοντας τις πιο παραδοσιακές ε, τράπεζες να προχωρήσουν σε καινοτομίες όσον αφορά το οικοσύστημα όπως το ονομάσατε. Και έπειτα, τι μέτρα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να περιορίσουμε τις τράπεζες σε ένα ποσοστό του ΑΕΠ της κάθε χώρας. Ξέρω ότι και εμείς κινδυνεύουμε πολύ όπως η Ισλανδία και η Ιρλανδία εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όμως έχουμε ένα οικονομικό κέντρο. Θα έπρεπε να μετριέται βάσει ενός ποσοστού του εθνικού ΑΕΠ, του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, μια που είμαστε ευρωπαϊκό οικονομικό κέντρο. Και για την ε, καθηγήτρια Λάτλεν. Είναι πάντα ενδιαφέρον να βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανταποκρίνεται με τα επιτόκια ε, σε σχέση με το τι κάνει το ΦΕΔ δηλαδή. Πολλές φορές είχε κατηγορηθεί ότι κρατούσε τα επιτόκια σε πολύ ψηλά επίπεδα. Παρ' όλα αυτά, ορισμένες χώρες της Ευρωζώνης δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από τη δημιουργία φούσκας. Οπότε μήπως δεν φτάνει αυτό το μέσο, τα επιτόκια δηλαδή, μήπως χρειάζονται και άλλα μέσα να έχει στη διαθεσή της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Όλες τώρα οι χώρες εκτός Ευρωζώνης δέχονται τώρα με τα κυκλικά μέτρα ότι πρέπει να έχουμε αύξηση των επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες εφόσον υπάρχει άνθεση της οικονομίας και μείωσή τους όταν υπάρχει ύφεση. Μήπως λοιπόν πρέπει να φροντίσει περισσότερο για τη σταθερότητα Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και όχι τόσο για ανάκαψη και άνθηση της οικονομίας όπως κάνει τώρα. Κύριε Χάτον, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Κοιτάξτε, είμαι υπέρ μιας εκδοχής που να ανταποκρίνεται περισσότερο στον 21ο αιώνα. Εγώ δεν βλέπω γιατί τα αποταμιευτικά ιδρύματα δεν μπορούν να κάνουν αυτά που λέτε. Με ρωτήσατε και κάτι άλλο για τις διάφορες κατηγορίες χρηματοοικονομικών παραγόγων. Έτσι όπως τίθεται όμως είναι λάθος το ερώτημα. Τι πιστεύουν οι τραπεζίτες ότι θα μπορούσε να γίνει που να είναι αποδεκτό για αυτό ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν. Όμως στην πραγματικότητα το ερώτημα πρέπει να είναι τι θέλουμε να κάνουν οι τράπεζες. Το έχουμε αποφασίσει πρέπει να έχουμε μια αρχιτεκτονική και να δούμε αν μπορούν να τη δεχτούν οι τράπεζες και έχουν αρκετό κέρδος. Έχουμε φτάσει σε κάποια όρια, όπως έδειξα και στις διαφάνειές μου, ακόμα και οι προσωπικές αμοιβέ. Οπότε δεν είναι δύσκολο γιατί οι τραπεζίτες θέλουν να κάνουν ε, όπως κάνουν τα πράγματα. Έτσι λοιπόν και ο επακεφαλής της Τράπεζας της Αγγλίας είπε πριν από δύο εβδομάδες ότι πρέπει οι μεγάλες τράπεζες να κοπούν σε κομμάτια. Η Ευρώπη λοιπόν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να το σκεφτεί αυτό. Οι Αμερικανοί το έκαναν σε ένα βαθμό λοιπόν, γιατί όχι εμείς. Να κοπούν σε κομμάτια αυτές οι μεγάλες τράπεζες, γιατί δεν εξυπηρετούν καμία λογική οικονομική λειτουργία. Να στηρίξουμε τις επενδύσεις. Ορισμένοι νομίζουν ότι θα είναι το τέλος του κόσμου. Όχι όμως τέτοια σκληρά ερωτήματα πρέπει να τα θέτουμε στους αυτούς μας. Μήπως αυτό πρέπει να γίνει. Ναι, όπως είπατε, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε ακούσει διάφορες επικρίσεις πριν από την κριση το 2000-2004 ότι κρατούσε τα επιτόκια πολύ ψηλά. Τότε οι τάσεις ήταν αποπληθωριστικές και γι' αυτό ανησυχούσε και το ΦΕΝΤΕ. Όμως πέρα από αυτό το θέμα που θέλει χωριστή συζήτηση, είναι αλήθεια και ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι για τα ίδια ονομαστικά επιτόκια υπήρχε πληθωρισμός σε μερικές περιπτώσεις για διαφορετικούς λόγους, είτε γιατί είχαν υπερβολική ανάπτυξη, αλλά πραγματικά επιτόκια είχαν πιο χαμηλά και αυτό είναι που έχει σημασία για τις φούσκες. Ισπανία και Ιρλανδία δηλαδή κύρια. Οπότε μπορούμε τη νομισματική μας πολιτική να την έχουμε σαν σύνολο ή πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ορισμένων χωρών. Έτσι κι αλλιώς όμως το θέμα των επιτοκίων όντως αντιμετωπίζει ορισμένα ζητήματα, όχι όλα. Συνεπώς, ένα επιτόκιο μπορεί να είναι συμβατό με πραγματικά επιτόκια σε ορισμένες περιπτώσεις. Ας πούμε στις Ηνωμένες Πολιτείες διαφέρουν τα επιτόκια στις πολιτείες μεταξύ τους εφόσον υπάρχουν ε, διαφορετικά ρυθμιστικά πλαίσια. Οπότε αν πάμε προς μια ευρωπαϊκή ρύθμιση αυτό δεν σημαίνει ότι διαφορετικές χώρες δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη ως διαφορετικές, εφόσον έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά, είναι όπως και με το θέμα των κύκλων. Λαμβάνουμε υπόψη μας διαφορετικές καταστάσεις, όπως αυτή την περίπτωση στην Ισπανία. Αν έρθουμε τώρα στο μέλλον των επιτοκίων την οικονομική σταθερότητα, εγώ έτσι τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας, και εδώ πιστεύω ότι τα επιτόκια πρέπει να αποτελούν μέσο για τον πληθωρισμό, για τον έλεγχο δηλαδή του πληθωρισμού. Αλλά από τη στιγμή που έχουμε φτάσει, εκεί που έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή, πρέπει να συμπληρώσουμε με άλλα μέσα, με μάκρο προληπτικά μέτρα από πλευρά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό είναι κάτι που χρειάζεται. Να σκεφτούμε προς αυτή την κατεύθυνση και μάλιστα γρήγορα. Ο κύριος Χάτον. πρέπει να πάρει το τρένο, οπότε οι δύο τελευταίες ερωτήσεις απευθύνονται σε εσά. Λοιπόν, Λίζα και Περβάνς, σας παρακαλώ γιατί πρέπει να έχουμε, έπρεπε να έχουμε περάσει το δεύτερο πάνελ. Δεν θα κάνετε ερώτηση, Ελίζα. Σύντομα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας. Ως ε, πανεπιστημιακός και εγώ θα ήθελα να σας ακούσω λίγο ακόμα. Έχουμε ένα στόχο, τον πληθωρισμό και έχουμε ένα μέσο που υποτίθεται ότι θα βοηθήσει την οικονομία είναι να ε, χαμηλώνουμε τα επιτόκια σε καιρούς ε, χαμηλής ανάπτυξης. Στη διάρκεια αυτής της κρίσης έχουμε αποκρινθεί πάρα πολύ και από την εντολή μας, τους κανόνες και από το να αντιμετωπίσουμε το, το πρόβλημα. Θυμάμαι πως υπήρχε μια εποχή που μειώνονταν ο ρυθμός ανάπτυξης και το ποσοστό ακόμα ανέβαινε από την Κεντρική Τράπεζα. Τι μαθήματα λοιπόν μπορούμε να αντλήσουμε εδώ πέρα, τι διδάγματα για την εντολή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για την νομισματική μας πολιτική. Και κανείς δεν μίλησε για τον ρόλο του Συμφώνου Σταθερότητας για να οδηγηθούμε ξανά σε ανάπτυξη. Θα ήθελα λοιπόν να επανέλθω στο πρώτο ερώτημα είναι διατεθειμένο το χρηματοπιστωτικό σύστημα να τροφοδοτήσει την οικονομία σε αντικυκλικό ρυθμό, στόχο. Αυτή είναι η ουσία. Αλλά τούτου λεχθέντος συμφωνώ πως ε, βράχει πρόθεσμα η δουλειά της ε, ΕΚΤ ήταν ε, σωστή, αλλά πρέπει να δούμε εδώ πέρα μέσω μακροπρόθεσμα τι γίνεται και ένα μέσο το οποίο δεν είναι μόνο βράχει πρόθεσμο, αλλά να βοηθήσει την οικονομία μακροπρόθεσμα. Θα ήθελα λοιπόν να δείτε έτσι λίγο αυτό το πλαίσιο. Ναι, είναι δύσκολο, δύσκολο να απαντήσω. Θέλω να επαναλάβω αυτό το οποίο είπα πριν. Νομίζω πως ο καθένας πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Η Κεντρική Τράπεζα, ξέρετε, κυρίως ασχολείται με τον πληθωρισμό. Τώρα είναι ανοιχτό το ζήτημα, το εάν η υπερβολική προσήλωση στον πληθωρισμό ήταν λάθος λόγω των ζητημάτων οικονομικής ε, αστάθειας. Τώρα η άλλη συζήτηση είναι η ανάπτυξη και ο ρόλος του Συμφώνου Σταθερότητας, αλλά εκεί πέρα το ερώτημα δεν πρέπει να απευθύνεται στους κεντρικούς τραπεζίτες, αλλά στο, στο πλαίσιο, στη συνθήκη. Ειδικά μετά την περίπτωση Ελλάδας, ε, τι διδάγματα αντλούμε και με βάση την περιορισμένη επιτυχία της Ευρωζώνης για να αντιμετωπίσει τα μακροπρόθεσμα ζητήματα, ανάπτυξη, τεχνολογία, καινοτομία κτλ. Αυτός δεν είναι ρόλος της Κεντρικής Τράπεζας. Αυτός είναι ο ρόλος ε, της ε, κυβέρνησης. Αλλά μπορούμε να σκεφτούμε αν ολόκληρη η συνθήκη διευκολύνει και δεν ε, εμποδίζει. Και θα έλεγα πως ε, αυτή είναι η στιγμή κατά την οποία πρέπει να σκεφτούμε γιατί ξέρετε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπαθούσε να στηρίξει το χρηματοπιστωτικό σύστημα μέσω εγγυήσεων, ε, ρευστότητας κτλ. Αλλά την περιόριζε η συνθήκη και σε περίοδους κρίσης Βεβαίως η δημοσιονομική πολιτική είναι πάρα πολύ σφιχτή, οπότε μπορούμε να έχουμε νομισματική πολιτική χωρίς να υπάρξει εμβάθυνση του δημοσιονομικού συντονισμού. Εγώ νομίζω όχι. Βεβαίω αυτά τα οποία λέω είναι οι ε, απόψεις μου αλλά νομίζω πως οι κανόνες συνθήκες πρέπει να αλλάξουν. Σας ευχαριστώ πολύ. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου πάνελ. Ε, θα ήθελα να ζητήσω από τα μέλη του δεύτερου πάνελ να έρθουν εδώ στο Προεδρείο. Σας ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας, τον χρόνο σας. Βεβαίως, αν θέλετε, μπορείτε να παραμείνετε. Αν θέλετε μπορείτε να, να παραμείνετε να καθίσετε εκεί. Uh, λοιπόν, έχουμε τώρα μαζί μας την κυρία Μαρία Ζαο από το Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο της Λισαβόνας και την κυρία Νίκολα Φούξ Χούντελν από το Πανεπιστήμιο Γκέτε. Δεν χρειάζεται να σας παρουσιάσω τα βιογραφικά τους. Πρώτα η κυρία Μαρία Ζαοροντρίγκες. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να, είναι έτοιμες οι διαφάνειές μου. Ήρθα εδώ για να σας μιλήσω για το εξής δύσκολο θέμα. Πώς μπορεί να δημιουργήσει η Ευρώπη νέες θέσεις απασχόλησης. Πρώτον, θα αναφερθώ στο εύρος της μόνιμης αυτής πρόκλησης που έχει η Ευρώπη και το δεύτερο είναι πού βρίσκονται ευκαιρίες για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Ένα τρίτο θέμα μου θα είναι μια πρόταση για απασχόληση και τέλος θα αναφερθώ στις πολιτικές προτεραιότητες που πρέπει να ακολουθήσουμε για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης. Θα ξεκινήσω με το, την ίδια την πρόκληση. Τα προβλήματά μας είναι δύο στην πραγματικότητα. Το ένα είναι η σχέση της απασχόλησης ή μάλλον της ανεργίας με την οικονομική ύφεση. Το άλλο είναι 10 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης. Ένα νούμερο δηλαδή. Στην ουσία μπορούμε να, να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε και μπορούσαμε 2005 με 2008 να δημιουργήσουμε 10 εκατομμύρια θέσει απασχόληση, τώρα μα τι χάνουμε εξαιτία τη ύφεση. Και προχωράμε σε ένα μέσο όρο 10% ανεργία. Αυτό λοιπόν από μόνο του είναι ένα πρόβλημα. Έχουμε όμως και ένα δεύτερο που μερικές φορές δεν αναφέρεται. Και αυτό είναι ο κίνδυνος της διαρθρωτικής ανεργίας. Δηλαδή η διάρθρωση της απασχόλησης αλλάζει στην Ευρώπη. Και πηγαίνουμε προς μια οικονομία βασισμένη στην γνώση. Φτιάχνουμε δηλαδή θέσεις απασχόλησης σε διαφορετικούς τομείς από ό,τι κατά το παρελθόν και δεν χρειαζόμαστε πια ε, το ίδιο είδος ανθρώπων για να απασχολήσουμε. Ίσως λοιπόν θα έπρεπε να επικεντρωθούμε στο δεύτερο. Και δέρχομαι σε ένα δεύτερο νούμερο. 70 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης θα ανοίξουν για νέες προσλήψεις. Και εδώ μιλάω για την καθαρή δημιουργία. Ε? Μιλάω για την απασχόληση που θα έπρεπε να υπάρχει, αλλά δυστυχώς δεν προορίζεται τόσο για του ανθρώπου που θα βρεθούν στην ανεργία και θα ψάχνουν καινούργια δουλειά τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, από τη μία μεριά έχουμε την ε, ανεργία εξαιτία τη ύφεση και το άλλο είναι η, λόγω της διάρθρωσης της απασχόλησης ανεργία. Δεν θα έπρεπε λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, να κοιτάξουμε το σημερινό ζήτημα. Κατά το παρελθόν, η πολιτική μας βασιζόταν στην προσφορά της απασχόλησης προκειμένου να προσελκύσουμε γυναίκες, νέους, νέους ανθρώπους στην αγορά εργασίας και η ευελιξία ασφάλεια στην αγορά εργασίας. Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι αυτά δεν πρόκειται να φτάσουν για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανεργίας στο μέλλον. Δεν φτάνουν για να έχουμε περισσότερη απασχόληση. Χρειάζονται μακροοικονομικές πολιτικές, καινοτομία και ένα δραστήριο ενεργό σύστημα διαβίου Άρα λοιπόν η προσοχή μας πρέπει να μετατοπιστεί και οι πολιτικές μας προτεραιότητες επίσης και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε εσείς οι ευρωβουλευτές ετοιμάζουμε επί του παρόντος την στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη δεκαετία και τη στρατηγική 2020. Άρα λοιπόν αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε τέτοιου είδους ζητήματα. Τώρα βέβαια θα μου πείτε πού θα βρούμε ευκαιρίες για νέες θέσεις απασχόλησης. Ε, λοιπόν, κατά κύριο λόγο, σε αυτού στους τέσσερις τομείς. Στις σφαιρικές αγορές και αναπτυγμένε χώρες, δηλαδή και αναπτυσσόμενες, αλλά βέβαια εξαρτώνται και από την παγκόσμια ανάκαμψη. Στις ευρωπαϊκές αγορές, οι οποίε πρέπει να είναι σε θέση να προσφέρουν νέε ευκαιρίες, αλλά και αυτό εξαρτάται από την ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά πόσο θα μπορέσουμε να εξελιχθούμε και Οικονομική και Νομισματική Ένωση κατά πόσο θα μπορέσει να συντονίσει ε, πολιτικές βάσει της νέας κατάστασης. Άρα με πολλά εάν και φόσον. Τρίτον, τρίτος χώρος που μπορεί να δημιουργήσει θέσει απασχόλησης είναι οι διάφορες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κοινωνία. Περιβάλλον, αλλαγές στο κλίμα, δηλαδή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά υγεία ε, καλύτερες υπηρεσίες για να στηριχθούν, για παράδειγμα, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Τέλος, στον τομέα της καινοτομίας και των νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Δεν μιλάμε μόνο για τη διαδικασία στην καινοτομία, αλλά μιλάμε και για τα προϊόντα το τελικό προϊόν. Μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης και καλύτερες θέσεις απασχόλησης. Αυτές είναι οι δυνατότητες που έχουμε. Αλλά πάντα βέβαια μιλάω για κάτι που είναι δυνητικά ικανό να δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Έρχομαι λοιπόν με τρεις συγκεκριμένες προτάσεις που πιστεύω ότι ταιριάζουν πάρα πολύ καλά με την στρατηγική μας για το 2020 που θέλει να προετοιμάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για μια πιο πράσινη οικονομία, για μια περισσότερο ευφύ οικονομία και για μια κοινωνία ε, στην οποία θα συμμετέχει όλος ο κόσμος και δεν θα αποκλείεται κανείς. Άρα λοιπόν πρέπει να φροντίσουμε να καταρτήσουμε τους ανθρώπους και να τους προσανατολίσουμε σε αυτά τα τρία είδη οικονομίας. Μια πιο πράσινη, περισσότερο ευθύ και μια οικονομία που θα φροντίζει ώστε να μην μένει στο περιθώριο κανείς στην κοινωνία. Όλα αυτά έχουν να κάνουν όμως και με νέους πόρους, νέους πόρους ενέργειας, για παράδειγμα. Πρέπει επίσης να φροντίσουμε να έχουμε και κατοικίες που να είναι περισσότερο οικολογικές, αλλά και οι μεταφορές μας πρέπει να είναι περισσότερο οικολογικές. Για την ευφύ οικονομία. Η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει σε αυτόν τον τομέα νέες θέσεις απασχόλησης. Πώς? Δημιουργώντας βιομηχανίες, επιχειρήσεις, και υπηρεσίες που να στηρίζουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Πριν από την κρίση, σε αυτό το τομέα δημιουργήθηκαν οι περισσότερες θέσεις απασχόλησης και αυτό μπορεί να γίνει και πάλι, εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Ο τρίτος τομέας τώρα που έχει να κάνει με την κοινωνία, μια κοινωνία που δεν θα αφήνει κανένα στο περιθώριο, αυτά έχουν να κάνουν με την ε, ε, μέρημνα για τα παιδιά, με την υγεία, με την εκπαίδευση και την κατάρτιση τελικά. Εδώ η Ευρώπη δυνητικά μπορεί να δημιουργήσει πολλές νέες θέσεις απασχόλησης. Έρχομαι τώρα στη μεθοδολογία. απαιτεί να χρησιμοποιήσουμε μια έννοια που είναι εταιρική σχέση για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε από κοινού μαζί καταρχήν την καινοτομία που είναι η κινητήρια δύναμη και την διαβίου κατάρτιση για να αποκτήσουν οι άνθρωποι τα προσόντα που χρειάζονται και τις δεξιοτεχνίες που χρειάζονται για τις νέες θέσεις απασχόλησης. Αυτό σήμερα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε επίπεδο κρατών μελών βρίσκεται σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Είναι αδύναμος κρίκος. Τι προτείνω δηλαδή. Πρέπει να ενισχύσουμε λοιπόν τις πολιτικές μας για την καινοτομία. Αλλά τι λείπει. Σήμερα έχουμε πολλά μέσα για την πολιτική μας, για την καινοτομία, τη βιομηχανική πολιτική, την έρευνα, αλλά όλα αυτά είναι κατακαιραματισμένα, δεν τα έχουμε βάλει μαζί. Για να πάρουμε σαν παράδειγμα την αυτοκινητοβιομηχανία. Υπάρχουν αυτά αλλά δεν συνδυάζονται μεταξύ τους. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν ευρωπαϊκές πλατφόρμες και αυτά τα μέσα να συνδυάζονται. Και σε εθνικό και σε περιφερειακό επίπεδο πρέπει να ενισχύσουμε αυτού του είδους ε, συνδυασμούς. Αλλά και πάλι η καινοτομία πρέπει να σχεδιάζεται όχι σαν μία πολιτική για μία ελίτ επιχειρήσεων ή περιφερειών ή ανθρώπων, όχι πρέπει να αφορά όλους τους ανθρώπους. Και δεν υπάρχει αυτό ακόμα. Βέβαια όλα θα εξαρτηθούν από τις αποφάσεις που θα ληφθούν εν ώψη της στρατηγικής 2020. Συγχρόνως, πρέπει να προχωρήσουμε και με την διαβίου κατάρτιση. Εγώ προτείνω το εξής. Δεν μας ενδιαφέρει μόνο να ανυψώσουμε το επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης αυξάνοντας το ποσοστό των Ευρωπαίων που θα έχουν διπλώματα δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας ε, εκπαίδευσης, αλλά το να τους εκπαιδεύσουμε στις κατάλληλες δεξιοτεχνίες και προσόντα. Και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με την διαβίω κατάρτιση. Δουλεύουμε πάνω σε μία πρόταση που μιλάει για ε, νέα προσόντα, για νέες θέσεις απασχόλησης. Τι σημαίνει αυτό. Εντοπίζουμε τις θέσεις απασχόλησης του μέλλοντος, που θα έχουμε δηλαδή στο μέλλον, ακριβώς για να μπορέσουμε να δούμε κάθε πολίτης που θέλει να προχωρήσει, με τι πρέπει να τον καταρτήσουμε για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις αυτών των νέων θέσεων απασχόλησης. Συχνά διαπιστώνουμε ότι δεν κάνουμε αυτό που πρέπει γιατί αυτό που πρέπει, αυτό που χρειάζεται είναι ένα πραγματικό σύστημα ευρωπαϊκό διαβίου κατάρτισης που να προσφέρει ευκαιρίες αλλά και ευκαιρίες για κάποιο είδους κινητικότητα στήλε Εράσμους. Ίσως να γνωρίζετε ήδη ότι μόνο το 1% των νέων έχουν πραγματικά την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το Εράσμος. Τέλος, τι οικονομικά μέσα διαθέτουμε. Γιατί βέβαια όλα αυτά που προτείνω θα είναι εφικτά μόνο εφόσον πρικοδοτηθούν από τα κατάλληλα οικονομικά μέσα, δηλαδή με κατάλληλα κονδύλια. Αν λάβουμε υπόψη μας τι πρόκληση μας περιμένει, για την απασχόληση δηλαδή, Χρειάζεται μια μακροοικονομική πολιτική υπέρ της ανάπτυξης. Και εδώ είμαστε σε ένα σταυροδρόμι, σε μια κρίσιμη καμπή. Από τη μια, το ΕΚΟΦΗΝ πηγαίνει προς την κατεύθυνση εξόδου από την κρίση μέσω φορολογικών πολιτικών. Από την άλλη μεριά έχουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το τελευταίο του Μαρτίου είπε ότι η οικονομική ενίσχυση πρέπει να συνεχιστεί μέχρι να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε ανάκαμψη. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να αποσύρουμε τα μέτρα ενίσχυσης παρά μόνο όταν αρχίσει η ανάκαμψη στην απασχόληση, όταν έχουμε νέες θέσεις απασχόλησης. Ένα δεύτερο θέμα είναι ο συντονισμός των οικονομικών μας πολιτικών. Δεν ε, πρέπει να αφήνουν απ' έξω την ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι και η φορολογική πολιτική αλλά και η εισοδηματική πολιτική πρέπει να συντονίζονται υπέρ μιας περισσότερο πράσινης και περισσότερο αφίους οικονομίας. Είμαστε μακριά όμως ακόμα από έναν τέτοιο συντονισμό. Δεν τον έχουμε. Τέλος πρέπει να αναπτύξουμε νέα οικονομικά μέσα. Εδώ δεν μιλά μόνο για καλύτερη χρήση των διευθυντικών ταμείων ή των κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Οικονο... Ε, Τράπεζας Επενδύσεων. Εδώ αναφέρομαι σε νέα μέσα. Ευρωμόλογα, για παράδειγμα και πάνω απ' όλα να φροντίσουμε ώστε το οικονομικό μας σύστημα θα μεταρρυθμιστεί έτσι ώστε να στηρίζει την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Βλέπετε ότι εδώ κάνω τη σύνδεση με αυτά που ακούσαμε στο πρώτο πάνελ, όχι μόνο από την Στέφανη Γκρίφιθ Jones, δηλαδή πρέπει να μεταρρυθμίσουμε το οικονομικό μας σύστημα έτσι ώστε τα χρήματα που έχουμε στη διάθεσή μας να στηρίζουν και την ανάπτυξη και την απασχόληση, αλλά και το πέρασμα σε μια πιο πράσινη οικονομία. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Φίξ Χιούντελ έχει τώρα το λόγο. Ευχαριστώ. Εγώ θα καλύψω τον ρόλο της αβεβαιότητας στην άμεση ανάκαμψη από την κρίση γιατί είναι ένας τομέας σημαντικός για τον οποίο δεν ξέρουμε ακόμα τι ρόλο μπορεί να παίξει η πολιτική και θα ήθελα μετά να αναφερθώ λίγο και στις μακροπρόθεσμες ε, στρατηγικές. Υπάρχουν λοιπόν δύο βασικά στοιχεία, δύο ερωτήματα. Πώς θα αυξηθεί η ζήτηση και πώς να αποφύγουμε την ανάκαμψη χωρίς δουλειές. Και εδώ πέρα βέβαια ε, υπάρχει πράγματι αβεβαιότητα και για τα δύο αυτά ζητήματα. Πράγματι η κρίση σήμαινε πως ε, είχαμε μείωση της ε, ζήτησης και ακολουθήσαμε την κεϊσιανή θεωρία που έλεγε πως οι κυβερνήσεις πρέπει να αυξήσουν την ζήτηση και οι περισσότερες πολιτικές αυτές ήταν επιτυχημένες. Υπήρχε επίσης συζήτηση για το εάν ε, η ζήτηση δεν υπάρχει σε κάποιες χώρες που έχουν υψηλά πλεονάσματα τρέχουσων συναλλαγών. Να δείτε λίγο εδώ πέρα τις ανισορροπίες τρέχουσων συναλλαγών. Βλέπετε πως η Γερμανία είναι η χώρα που έχει οπωσδήποτε το μεγαλύτερο πλεόνασμα τρέχουσων συναλλαγών. Οπότε η τοπική ζήτηση, αν θέλετε, έχει πέσει. είναι ένα πλεόνασμα αυτό εις βάρος του υπόλοιπου κόσμου, εις βάρος των υπολείπων κρατών μελών. Βλέπετε ένα παρόμοιο γράφημα σε σχέ... των ε, κρατών μελών της Ένωσης μεταξύ τους και τώρα το βλέπετε ως ποσοστό του ΑΕΠ. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το διαβάσετε. Βλέπετε εδώ πέρα η Ολλανδία έχει ως ποσοστό του ΑΕΠ το υψηλότερο πλεόνασμα, γιατί ως ποσοστό του ΑΕΠ η Γερμανία δεν έχει τόσο μεγάλο πλεόνασμα. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν ελλείμματα και άλλες που έχουν πλεονάσματα, οπότε μπορεί να αυξηθεί κάποια η τοπική ζήτηση. Οπότε, πώς μπορούμε να αυξήσουμε την ζήτηση. Φανταστείτε πως αυξάνεται η ανάπτυξη και οι περισσότεροι θεωρούν πως θα έχουμε θετική ανάπτυξη φέτος, αυξάνουν οι μισθοί και θεωρούν όλοι πως αυτομάτως θα αυξηθεί και η ζήτηση. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, θεωρώ εγώ. Δεν έχουμε αρκετή έρευνα επ' αυτού. Να σας δείξω λίγο μια καθημαϊκή έρευνα από τον σχετική νομοθεσία του 2008 στη ΣΥΠΑ όταν έστειλαν την επιστροφή της εφορίας στα νοικοκυριά μεταξύ κάτι, ε, επιταγές μεταξύ 300 και 2.000 δολαρίων ανά νοικοκυριό και αναμένονταν πώς θα τα ξοδέψουν αυτά, αλλά μόνο 20% των νοικοκυριών είπαν πώς θα τα ξοδέψουν αυτά. Τα περισσότερα νοικοκυριά σε καιρούς κρίσης όταν έχουν περισσότερα χρήματα τα αποταμιεύουν ή αποπληρώνουν το χρέος, που και αυτό είναι ένα είδος αποταμίευσης. Κάτι το οποίο μας προξενεί ακόμη ε, μεγαλύτερη έκπληξη είναι πως τα πιο πλούσια και τα πιο γερασμένα νοικοκυριά λένε πως θα τα ξοδέψουν. Και αυτό μας προξενεί η έκπληξη, γιατί θεωρούσαμε πως τα νέα και φτωχά νοικοκυριά βεβαίως θα αυξαναν τη ζήτηση, αλλά τα στοιχεία μας δείχνουν το αντίθετο. Τι συμβαίνει λοιπόν. Η αβεβαιότητα παίζει μεγάλο ρόλο η δική μου έρευνα βρήκε πως ε, υπάρχουν προληπτικές αν θέλετε αποταμιεύσεις για να προστατευτεί κανείς από τις μελλοντικέ διακυμάνσεις του εισοδήματος. Και τι συνέβη εδώ πέρα. Η αβεβαιότητα των οικοκυριών αυξήθηκε, κάτι το οποίο ισχύει ιδιαίτερα για τα νεαρά νοικοκυριά που δεν ξέρουν τι θα γίνει ακόμα στην αγορά εργασίας και βεβαίως χάθηκαν και θέσεις εργασίας ε, και αυτό έπληξε κατά κανόνα τα φτωχά νοικοκυριά. Οπότε υπάρχει μια γενικότερη αβεβαιότητα για το πώς θα λάβει η χώρα η ανάκαμψη, αν θα έχουμε ξανά μια ύφεση, διπλή ύφεση ή αν θα έχει σχήμα Y ε ε, ή οτιδήποτε άλλο. όσο υπάρχει αυτή η αβεβαιότητα, ακόμα και αν αρχίζει να αυξάνεται το ΑΕΠ και η μισθή, δεν σημαίνει πως θα ακολουθεί συζήτηση. Μία άλλη ψυχολογική αβεβαιότητα, την οποία θέλω να αναφέρω, είναι το θέμα της εμπιστοσύνης. Υπάρχει επίσης ε, έρευνα στο μικρο και στο μάκρο επίπεδο που δείχνει πως η εμπιστοσύνη είναι μεγάλη. Ε, έχει μεγάλη σημασία και μεταξύ χωρών και μεταξύ ανθρώπων ε, δηλαδή. Και βλέπετε τη σχέση με το ΑΕΠ. Χώρε με υψηλότερο ποσοστό εμπιστοσύνη έχουν και υψηλότερο ΑΕΠ. Χώρες οι οποίες εμπιστεύονται περισσότερο η μία την άλλη μεταξύ του ε, έχουν και μεγαλύτερο όγκο εμπορίου μεταξύ του. και αυτό το οποίο ακούμε τώρα συνέχεια είναι πως η κρίση κατέστρεψε την εμπιστοσύνη στο οικονομικό σύστημα. Ένα νέο χαρακτηριστικό αυτή τη κρίση εάν τη συγκρίνουμε με παλαιότερες υφέσεις. Και δεν νομίζω ότι ξέρουμε πάρα πολύ καλά σε τι θα μας οδηγήσει αυτό όσον αφορά τη συμπεριφορά εταιριών και νοικοκυριών. Επίσης βλέπουμε πώς καταστρέφεται η εμπιστοσύνη μεταξύ ανθρώπων και στις οικονομικές συναλλαγές και είναι σαφές πως οι προτιμήσεις και η συμπεριφορά των ανθρώπων διαμορφώνεται από την οικονομική εμπειρία που είχαν. Π.χ. αν δούμε τη μακροπρόθεσμη εμπειρία, οι άνθρωποι στην Ανατολική Γερμανία έχουν την εμπειρία του κομμουνισμού, αλλά αυτό ισχύει και σχέση με τη βραχυπρόθεσμη εμπειρία. Άλλη ε, έρευνα δείχνει πως ανάλογα με την εμπειρία και αν είχαν κέρδη ή όχι στις χρηματαγορές είναι διατεθειμένοι να αναλάβουν κινδύνους ή όχι. Οπότε, ε, τι ακόμα δεν ξέρουμε ποιες είναι οι συνέπειες αυτής της εμπιστοσύνης που χάθηκε. το δεύτερο σημείο που θέλω να αναφέρω. Πρέπει να φοβόμαστε μία ανάκαμψη χωρίς δουλειές, κάτι το οποίο είχαμε στις ε, δύο τελευταίες υφέσεις της ΕΠΑ, που αυξήθηκε το ΑΕΠ, αλλά δεν αυξήθηκαν οι δουλειές. Οι μειώνονταν ε, κιόλα για κάποιον καιρό και χρειάστηκαν δυόμιση χρόνια για να φτάσουν οι θέσεις εργασίας στο ίδιο επίπεδο με αυτό που είχαν πριν την ύφεση και οπωσδήποτε αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικέ θεωρίε για το γιατί οδήγησε σε αυτή την ανάκαμψη χωρίς ε, δουλειές. Μία θεωρία λέει πως υπήρχε μία ανακατανομή ή ότι οι θέσεις ήταν σχετικά ρηχές και δεν δημιουργήθηκαν νέες θέσεις εργασίας αλλά αυξήθηκαν τα ωράρια. Τόσο αυτή η κρίση δεν ήταν ρηχή και σύντομη αλλά βλέπουμε πως αυξήθηκε η αβεβαιότητα των επιχειρήσεων και βεβαίως ε, σε αυτή την περίπτωση περιμένουν οι επιχειρήσεις ε, αντί να δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας. Και εδώ πέρα σε αυτό το διάγραμμα βλέπετε το αρνητικό αποτέλεσμα της αβεβαιότητας στην παραγωγή που κρατάει αρκετά μεγάλο διάστημα. Τι έγινε λοιπόν στην τωρινή κρίση με την αβεβαιότητα. Αυτό είναι ένα δείκτης από τη Γερμανία, ο δείκτης Ήφο, τον έχετε ξανακούσει ίσω αφορά την εμπιστοσύνη, την αισιοδοξία των επιχειρήσεων. Βλέπετε στο τέλος του διαγράμματο είναι σαφές πω η αβεβαιότητα αυξήθηκε κατά πολύ κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτή είναι η αβεβαιότητα των επιχειρήσεων για το τι θα κάνει η οικονομία και για το τι θα κάνει η δική του η επιχείρηση. Αν οι θα είναι θετικέ ή αρνητικές. Συμπερασματικά λοιπόν θα έλεγα πως η αβεβαιότητα και η εμπιστοσύνη είναι σημαντικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά που έχουν οικονομικό αντίκτυπο και δεν είναι σαφές ακόμα το τι μπορεί να κάνει η πολιτική για να αυξήσει την βεβαιότητα και την εμπιστοσύνη αλλά σκεπτόμενη την κρίση την τρέχουσα κάποια μέτρα είναι ε, σαφή Οπότε οτιδήποτε αυξάνει την αβεβαιότητα επιχειρήσεων και νοικοκυριών πρέπει να αποφθεί και όπως είπαν και οι περισσότεροι συναδελφοί μου ήδη, θα έλεγα και εγώ πως μια αργή στρατηγική εξόδου για το πώς θα καταργηθούν σταδιακά οι α, πολιτικές αυτές είναι σημαντική οπότε ε, να έχουν εμπιστοσύνη νοικοκυριά και επιχειρήσεις ε, στην ε, πολιτική αυτή, ότι θα συνεχιστεί δηλαδή μέχρι να ανακάμψει η οικονομία. Και τέλος, συντονισμός σε κάποια μέτρα πολιτικής σε ευρωπαϊκό επέδο θα μπορέσει οπωσδήποτε να βοηθήσει γιατί θα δημιουργήσει ένα σαφές πλαίσιο των κοινών στόχων, των κοινών πολιτικών για να καθοδηγηθούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Τέλος λοιπόν να μιλήσω δύο λεπτάκια για τη μακροπρόθεσμη στρατηγική και εδώ πέρα συμφωνώ με τα υπόλοιπα μέλη του πάνελ πως οπωσδήποτε όσον αφορά τη μακροπρόθεσμη στρατηγική υπάρχουν κάποια ακόμα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Η Ευρώπη έχει συγκριτικό πλεονέκτημα στην έρευνα και ανάπτυξη και θα πρέπει να δοθεί άρα βάρος στις δεξιότητες και στην έρευνα. Αν δούμε λοιπόν τώρα Δαπάνε έρευνα και ανάπτυξη βλέπετε πω υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφοροποίηση και βλέπετε πώ δεν έχουν φτάσει όλοι το 3% που θέλει να θέσει ω το 2020 στόχο η Κομισιόν και να πω επίση πω δεν είναι όλε οι δαπάνε ίδιε, οπότε πρέπει να ξαναδούμε το πω γίνεται η έρευνα και ανάπτυξη εγώ θεωρώ πως πρασινε τεχνολογιε θα πρέπει να παίξουν σημαντικό ρόλο γιατί έχουμε ένα ε, συγκριτικό πλεονέκτημα. Εδώ πέρα είναι προωθημένο το οικολογικό κίνημα. Θα γίνει πιο σημαντικό και στην Κίνα και στην Ινδία. Οπότε πρέπει να, ε, εάν μπορέσουμε να τους δώσουμε εμείς τεχνολογίες, έχουμε μια ευκαιρία ανάπτυξης. Τέλος, δαπάνες εκπαίδευσης, η μπλε στήλη είναι ποσοστό του ΑΕΠ, και δεξιά έχουμε σύγκριση με ΙΠΑ, Ελβετία και τα λοιπά, αλλά και εδώ πέρα δεν είναι μόνο χρήματα, πρέπει να σκεφτούμε πού θα τα διοχετεύσουμε. Και μία τελευταία παρατήρηση στη Γερμανία γνωρίζω πως ε, ε, πάνω από τις μισές φοιτήτριες είναι γυναίκες αλλά μετά μένουν πίσω στην αγορά εργασίας γιατί είναι και προσωπικό το ζήτημα, αλλά υπάρχουν και κοινωνικές ε, θετικές επιπτώσεις. Βλέπετε εδώ πέρα την συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι πολύ πιο κάτω από το 57% που θέλει η Κομισιόν. Ε, βλέπετε τι γίνεται εδώ πέρα και μητέρες με παιδιά ακόμη χαμηλότερο. Οπότε πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι πόροι που υπάρχουν στην κοινωνία με το να μπουν οι γυναίκες στην αγορά εργασία. Uh, τι μπορεί να κάνει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σαφές πως μια συντονισμένη ευρωπαϊκή πολιτική θα βοηθήσει ειδικά εκεί όπου υπάρχει ήδη ολοκλήρωση. Ακούσαμε σήμερα πάρα πολλά για τις ε, χρηματαγορές, τη ρύθμισή τους. Ναι, αλλά πρέπει να υπάρχει και συντονισμός. Ε, εκεί πρέπει να προωθηθεί η ολοκλήρωση, π.χ. στην αγορά εργασίας που ακόμα είναι αρκετά χαμηλή στην Ευρώπη. Δεδομένου το ότι επί της ε, αρχής υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση των εργαζομένων. Μπορούμε επίσης να δούμε τις βέλτιστες πρακτικές. Γιατί η συμμετοχή των μητέρων στην αγορά εργασίας είναι πολύ ψηλότερη σε άλλες χώρες, σε κάποιες χώρες. Και μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και να τα συζητήσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά αυτό το οποίο αναφέρθηκε νομίζω είναι η καινοτομία και πώς θα οθήσουμε την ατομική πρωτοβουλία. Αυτό είναι δύσκολο. Πρέπει να ε, είναι σαφές πως πολλά πράγματα θα οθησουμε την ατομικη πρωτοβουλια αυτο ειναι δυσκολο πρεπει να ειναι σαφες πως πολλα πραγματα θα σε περιφερειακό επίπεδο και δεν βοηθάει πάντα ο συντονισμός. Αλλά ε, εντάξει. Γενικά νομίζω πως υπάρχει εδώ πέρα αρκετό περιθώριο ευρωπαϊκής πολιτικής. Ε, Ευχαριστώ και εγώ πολύ, ο Και τώρα καλώ τους συναδέλφους Α, ποιος θα ρωτήσει πρώτος. Η Ελίζα. Ευχαριστώ και τις δύο μιλήτριες. Ήταν μεγάλο ενδιαφέρον ε, τα γραφήματα της τελευταίας ομιλήτριας. Μπορείτε να πάτε πίσω στην ε, πρώτη διαφάνεια παρακαλώ. Αξίζει σχολιασμού. πρέπει να, το, να την αναλύσουμε αυτή την διαφάνεια πολύ προσεκτικά. Κοιτάξτε τι συμβαίνει. Όταν την κοίταζα, τη στιγμή που διέτρεχα άλλα χαρτιά ε, και ξαφνικά ε, σήκωσα το κεφάλι, νόμιζα ότι αυτή η μακριά γραμμή, ε, αυτό το, το μεγάλο πλεόνασμα ήταν της Κίνας. Αλλά δεν είναι έτσι. Όταν έχουμε τόσο δειλή ανάκαμψη στην Ευρώπη, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τελικά. Γιατί αυτή η δειλή ανάκαμψη και η υπερβολική συγκέντρωση εξαγωγών στην εσωτερική αγορά, δηλαδή οι χώρες εξάγουν μεταξύ τους, η μία στην άλλη. Τελικά που καταλήγουμε. Πολύ φυσικά, πολύ λογικά, σε ένα πολύ αυστηρό και βίο ανταγωνισμό. Τελικά λοιπόν δημιουργήσαμε ένα μοντέλο στην Ευρώπη όπου έχουμε ε, πλεονάσματα στη Γερμανία και στις βόρειες οικονομίες και έχουμε ελλείμματα σε όλες τις υπόλοιπες οικονομίες. Και αυτό δεν μπορούμε να το εμποδίσουμε. Γιατί εδώ πέρα αυτό συνδέεται και με την ε, εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη στην Ευρώπη και στην ευρωπαϊκή αγορά. Και τελικά αυτό είναι ένα ατελέσφορο παιχνίδι. Κάπου πρέπει να διδαχθούμε από όλη αυτή την ιστορία, γιατί να το συνδυάσουμε με τις διαφορές του ΑΕΠ, τις, τις διαφορές του κατακεφαλήν ΑΕΠ αναοικονομία, καταλαβαίνουμε ότι κάθε χρόνο τελικά να παράγουμε αυτό το μοντέλο. Και αν το συνδυάσουμε αυτό με το πακέτο σταθερότητας και ανάπτυξης, η κατάσταση γίνεται εκρηκτική τελικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό λοιπόν τονίζω με μεγάλη ένταση το τρόπο που μπορούμε να αναπτυχθούμε βιώσιμα, να δημιουργήσουμε θέσεις απασχόλησης, να λάβουμε υπόψη το περιβάλλον. Πρέπει να βρούμε μία λύση για αυτό το θέμα. Αυτό το άλμα από την μακροοικονομική ε, κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε τώρα σε ένα άλλο είδους ανάπτυξη είναι το μεγάλο ερωτηματικό. Ε, σε γενικό επίπεδο έχουμε ανάπτυξη 1%. Αλλά έχουμε πολλές διαφορές από χώρα σε χώρα. Το 1% είναι ο τελικός μας όρος. Το 1% ανάπτυξη δημιουργεί ανεργία κάθε χρόνο. Ε, θέλουμε ανάπτυξη πάνω από 2% για να έχουμε θέση απασχόλησης. Μέχρι να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα έχουμε πρόβλημα. Το θέμα είναι πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Πώς μπορούμε να φτάσουμε σε επίπεδα ανά, ανάπτυξης. Είμαστε σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, σε ένα παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Πώς μπορεί η Ευρώπη να αναπτυχθεί στα πλαίσια μιας παγκόσμιας οικονομίας. Τελειώνω, τελειώνω, Πρόεδρε. Αυτό τώρα μας παραπέμπει στη στρατηγική του 2020. Υπάρχουν δύο-τρεις καινοτομίες στην ε, στρατηγική και κάποια παλιά πράγματα. Η καινοτομία ποια είναι προσπαθεί να αντιμετωπίσει μια εξωτερική ατζέντα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Χρειαζόμαστε αυτό το άνοιγμα, γιατί αλλιώς θα κολλήσουμε στην ανάπτυξη του 1%. Δεύτερον, οι βιομηχανικές πολιτικές για πρώτη φορά ξαναθέτουμε στο πλαίσιο στην εξίσωση τις βιομηχανικές πολιτικές. Αλλά αυτό που δεν αντιμετωπίζουμε είναι τα μέσα, τα εργαλεία για να εφαρμόσουμε τη στρατηγική και ο δεύτερος άγνωστος χ στην εξίσωση είναι η σύγκληση. Είναι τεράστιο θέμα αν θέλουμε να δούμε τι μας έδωσε η παλιά ατζέντα της Λισαβόνας. Αν δεν αντιμετωπίσουμε τα, τα προβλήματα της Λισαβόνας, ε, αναπαράγουμε αυτές τις ανισορροπίες. Πρόεδρος, πριν δώσω το λόγο στις δύο κυρίες, θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να μην παραβλέπετε τις άλλες διαφάνειες Παραδείγματο χάρη το πλεόνασμα των εξαγωγών σε σχέση με το ΑΕΠ. Εκεί ήταν πρώτη η Ολλανδία και μετά η Γερμανία, 30%. Και εν συνεχεία το άλλο γράφημα που μιλάει για τις εξαγωγές στην Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Η Γερμανία ήταν πολύ κατώτερη εκεί. Δεν πρέπει να βλέπετε μονόπαντα το θέμα αυτό, δηλαδή μόνο το γράφημα αυτό στο οποίο εστιάσατε. Πρέπει να δείτε όλη την εικόνα. Ναι, Όντω, θα πρέπει να είναι τα πράγματα όχι απόλυτα, αλλά σχετικά. Αν υπολογίσουμε όμω ε, το εμπορικό πλεόνασμα ή έλλεισμα σε σχέση με το ΑΕΠ, τελικά να παράγουμε τα ίδια μοντέλα. Στο δεύτερο γράφημα έχουμε το ποσοστό του ΑΕΠ. Αν έχουμε υψηλότατο ΑΕΠ. Κοιτάξτε, εγώ δεν, ε, δεν μιλάω εναντίον κανενός και καμία ιδέα. Αλλά αν ομφαλοσκοπούμε στο εσωτερικό της ε, εσωτερικής αγοράς κάποιοι κερδίζουν και κάποιοι χάνουν μέσα στην Ευρώπη. Δεν κερδίζουν όλοι. Και εγώ θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπε ο Πρόεδρος, λέει η κυρία Φούξ ε, Σούντελ. Φυσικά τα απόλυτα μεγέθη έχουν σημασία. Φυσικά αν είσαστε μεγάλη χώρα η ζήτησή σας έχει μεγαλύτερη σημασία από ότι αν είσαστε μικρή χώρα. Αν δείτε όμως αυτό το γράφημα σε σχέση με, με το ποσοστό του ΑΕΠ θα δείτε ότι το γερμανικό πλεόνασμα είναι σχετικά μικρό, είναι 5%. Είναι σημαντικό, εντάξει, αλλά δεν είναι ακραίο, δεν είναι υπερβολικό. Δεν μοιάζει με τη Κίνας, ας πούμε, ούτε κατά διάνοια. Ε, το πλεόνασμα επίσης ε, προκύπτει και από τις ε, πολιτικές σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Σε ορισμένε περιόδους μπορούμε να έχουμε πλεόνασμα και σε άλλες έλλειμμα. Υπάρχει, υπάρχουν αποχρόντες λόγοι γι' αυτό. Από την άλλη συμφωνώ μαζί σας ότι υπάρχει ανομοιογένεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ορισμένες χώρες έχουν μεγάλα πλεονέσματα και άλλες μικρές ε, μεγάλα ελλείμματα. Γι' αυτό ακριβώ είναι δύσκολο σε ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε συντονισμένε πολιτικέ που είναι κατάλληλε για όλε τι οικονομίε. Με αυτή την έννοια είναι δύσκολο για την Ευρώπη να αντιμετωπίσει αυτή την ε, ανομοιογενή κατάσταση στα κράτη-μέλη. Αλλά μην νομίζετε ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι μηδέν πηλίκον. Όλοι αποφελούνται από το εμπόριο. Φυσικά θα υπάρχουν ε, περίοδοι όπου κάποιες ε, χώρες εξάγουν περισσότερο από κάποιες άλλες κτλ. Και έχετε δίκιο ότι αυτή η κατάσταση υπάρχει εδώ και καιρό. Θα πρέπει να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε, τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, αν είναι βιώσιμη η κατάσταση ή όχι. Αλλά δεν είναι καταστροφική. Αυτό μπορώ να πω σε τελική ανάλυση. Ε, πάντως, για το συντονισμό των πολιτικών μας, αυτό το ζήτημα αποτελεί πραγματική πρόκληση. Είναι κεντρικό αυτό το θέμα. Η δική μου αξιολόγηση για τη στρατηγική για το 2020, ε, όπως είναι αυτή τη στιγμή, γιατί είναι ούτως ή άλλως υποσυζήτηση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, είναι ότι αν θέσουμε το ερώτημα πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η στρατηγική αυτή του 2020 θα είναι πιο αποτελεσματική από τη στρατηγική της Λισαβόνας, πώς θα εξασφαλίσουμε ότι διδαχτήκαμε τα μαθήματα της Λισαβόνας, Μπορούμε να πούμε το εξή. Με τι προτάσει που έχουμε επιτάπητο, η δική μου τουλάχιστον εκτίμηση είναι ότι μα λείπουν τα μέσα και τα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε δύο προβλήματα. Πρώτον, να επιταχύνουμε τη μετάβαση προς μια πράσινη και έξυπνη οικονομία που συμπεριλαμβάνει όλους. Αυτό για να γίνει θέλει πολιτικά ισχυρά μέσα και χρηματοπιστωτικά ισχυρά μέσα. Υπάρχει όμως και ένα δεύτερο θέμα. Το θέμα της διαφοροποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της ανομοιογένειας στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να εντοπίσουμε τα εργαλεία για να υπάρχει μεγαλύτερη σύγκληση προς αυτούς τους κοινούς στόχους. Αν θέλουμε να κινηθούμε μαζί προς μια πράσινη, πιο πράσινη και πιο έξυπνη οικονομία, θέλουμε μέσα για τη σύγκληση. Αν δούμε τα συμπεράσματα του τελευταίου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η τελευταία μέρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, προσθέθηκε τελευταία, ε, προσθέθηκε η λέξη σύγκληση. Τώρα υποτίθεται ότι θα πρέπει να βρούμε ένα πλαίσιο για την ε, εποπτεία και για πρώτη φορά ψάχνουμε όχι μόνο την ανάπτυξη, τα ελλείμματα, αλλά και της ε, ισορροπίας των εμπορικών ισοζυγίων και το, της την ανισορροπία ή όχι του ισοζυγίου τρέχουσων πληρωμών. Ψάχνουμε ένα πιο συνεκτικό, ένα πιο πλήρες πλαίσιο για να προχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά έχω να πω εγώ. Ευχαριστώ. Το κύριο θετικό που έχει η Ευρώπη είναι η εσωτερική της αγορά. Είναι το ατού και κανείς δεν το είπε αυτό. Εφόσον λειτουργεί η εσωτερική αγορά, θα έχουμε και ανάκαμψη. Είναι η μεγαλύτερη αγορά του κόσμου η ευρωπαϊκή αγορά. Και ο κύριος Μόντι ετοιμάζει κάτι σχετικά. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Μαρία Ζαροντρίγκες. Εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να κατέψουμε τις πληγές της εσωτερικής αγοράς. Και για την ε, κυρία Φουξούντερτ. Και εκείνη το ανέφερε. Αυτό που ο Μπιλ Κλίντον βασικά είπε ότι η οικονομία αυτή είναι η ανόητη και όχι άνθρωπος. Στους Financial Times διάβασα ότι μία σημαντική υψηλού επίπεδου διάσκεψη που έκανε ο κύριος Σόρος, οργάνωσε ο κύριος Σόρος, είπε ότι τελικά η ψυχολογία, ο άνθρωπος είναι κάτι πολύ πιο σημαντικό από τα νούμερα. Εσείς τι λέτε για το θέμα αυτό του σεμιναρίου του κύριου Σόρος. Κοιτάξτε, για, την, ε, για το θέμα αυτό. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μια καλή ιδέα. Ένα καλό σημείο εκκίνηση. Ότι έτσι κι αλλιώ για την ενιαία αγορά χρειαζόμαστε ένα συμβιβασμό. Πρέπει να πάμε περισσότερο σε βάθο όσον αφορά τι ευκαιρίε που δίνει η εσωτερική αγορά, αλλά αυτέ τι ευκαιρίε πρέπει συγχρόνω και να τι συνδυάσουμε με κάποιε προποθέσει. Σύγκληση προ κοινέ προδιαγραφέ και σε κοινωνικό επίπεδο και σε περιβαλλοντικό επίπεδο και φορολογικά. Και γι' αυτό το τελευταίο, εγώ δεν μιλάω για αναρμόνιση, εντάξει, μιλάω για ένα ζωτικό θέμα που θα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό είναι ότι αργά ή γρήγορα όλες οι κυβερνήσεις θα αναγκαστούν να αυξήσουν τους φόρους. Εδώ λοιπόν πρέπει να πάμε προς μία ενιαία κατεύθυνση αναγκαία για την ανάκαμψη που είναι όπως και να έχουν τα πράγματα δεν πρέπει να αυξήσουμε το άχθος της εργασίας. Να κατευθυνθούμε αλλού. Ε, περιβαλλοντικός φόρος, ε, φόρος στις οικονομικές συναλλαγές, αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε συντονισμένα αν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Συνεπώς δεν ξέρουμε ακόμα, περιμένουμε την έκθεση του Μόντι. Πάντως υπάρχει άμεση διασύνδεση ανάμεσα στο να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που δίνει η νέα αγορά από τη μία, αλλά από την άλλη να συντονίσουμε τις δημοσιονομικές και φορολογικές μας πολιτικές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζω ότι η έκθεση του Μότι θα καταλήξει στο ίδιο συμπέρασμα. Τώρα κάτι άλλο δεν είμαι σίγουρη αν σας κατάλαβα καλά. Ο κύριος Σόρος το δότησε μία πρωτοβουλία για εναλλακτικέ λύσεις στην οικονομία ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε κρίσεις όχι μόνο σε και που μόλις περάσαμε αλλά και σε επόμενες. Διάβασα λοιπόν τα μέσα ενημέρωσης είπαν ότι δεν υπήρξε συνένεση, εντάξει αυτό δεν είναι και δύσκολο γιατί υπάρχουν φυσικά διαφορετικές απόψεις και τάσεις, όμως υπήρξε αναγνώριση για το ότι πρέπει να υπάρξει ένας πιο στάνταρ τρόπος σκέψης στα οικονομικά για να ξεπερνάμε τέτοιες κρίσεις. Πώς είναι περίπλοκο. Γιατί βλέπουμε ότι η κενησιακή θεωρία επιστρέφει και άλλες σχολές. Όμως δεν έχουμε καταλήξει σε μία συνθετική άποψη που να είναι αξιόπιστη. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τη συζήτηση σε βάθος. Γιατί η κλασική σχολή σκέψης είναι ξεκάθαρη, αλλά χρειαζόμαστε και άλλες εναλλακτικές. Έχω ένα κατάλογο μιλητών με τέσσερις ακόμα. Ο χρόνος όμως περνάει. Ίσως ε, να μην ε, επιμείνουμε περισσότερο. Περβάν στο τέλος θα πάρεις εσύ το λόγο. Εγώ τώρα τι έχω σημειώσει εδώ. Θέλω να ρωτήσω και τις δυο σας το εξής, κύριε Ροντρίκη, εσείς πρώτα. Έχουμε δύο εξελίξεις που επηρεάζουν την αγορά εργασίας είναι οι δημογραφικές εξελίξεις και το γεγονός ότι έχουμε όλο και περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι σταματάνε τις σπουδέ τους. Που σημαίνει ότι έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε αρκετούς καταρτισμένους στο επίπεδο που θέλουμε, αλλά και από αυτούς που προχωράνε εγκαταλείπουν κάποια στιγμή. Στην Γερμανία είναι της τάξης του 15%, στους 7. Ανησυχητικό στοιχείο. Αναρωτιέμαι λοιπόν, αφού είναι έτσι τα πράγματα, δεν θα έπρεπε να επιταχύνουμε κάπως τις προσπάθειές μας για να δημιουργήσουμε μια πραγματικά ευρωπαϊκή αγορά εργασίας που δεν την έχουμε. Προσπαθούμε να ολοκληρώσουμε την εσωτερική αγορά, χωρίς να έχουμε όμως μια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Λοιπόν, συμφωνείτε με αυτό. Και δεύτερον, η διαδικασία της Μπολόνια πιστεύετε ότι μας βοηθάει να δημιουργήσουμε τις δεξιοτεχνίες που θα χρειαστούμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι η διαδικασία της Μπολόνια διδάσκει κάποιες δεξιοτεχνίες, αλλά χωρίς όμως να έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Ενώ χρειαζόμαστε πραγματικά όριμες και αυτόνομες, αυθύπαρκτες προσωπικότητες και αυτό δεν το κάνει η διαδικασία της Μπολόνια. Κάτι άλλο τώρα στα γερμανικά προς την ε, κυρία Φούξ Σιντελν. Μιλήσατε για την ε, εμπιστοσύνη η οποία επλήγει. Συμφωνώ. Το ερώτημά μου είναι έχετε εμπειρικά δεδομένα αποδείξεις για το ότι αύξησε την μαύρη οικονομία αυτή η χαμένη εμπιστοσύνη, είτε αύξησε τη διαφορά, και άλλα τέτοια φαινόμενα που δεν χρειαζόμαστε στην σημερινή μας κατάσταση. Ευχαριστώ. I have you on the list. Ναι, ναι. και εσείς στον κατάλογο. Η κυρία Μπέρες. Μια που δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Μήπως να ακουστούν πρώτα οι ερωτήσεις και μετά να απαντήσουν οι προσκεκλημένες μας. Μα κύριε Τόμσον, είσαστε στον κατάλογο. Καλά καλά εντάξει αφού συμφωνείτε περνάμε στη κυρία Γκέπαρτ που είναι η επόμενη ομιλήτρια, μετά η κυρία Ουλμάγερ και μετά η κυρία Τόμσον. Και μετά η Περβάνς βέβαια. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με ένα από τα ερωτήματα του κύριου Κλίντς. Την λέξη κλειδί εμπιστοσύνη που αναφέρθηκε. Εάν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στο μέλλον του ανθρώπου, ε, όχι μόνο δεν θα ξοδέψει, αντιλαμβάνεσαι τι θα γίνει. Αυτή ακριβώς είναι η αποστολή της πολιτικής να δημιουργήσει μια εμπιστοσύνη για να αρχίσουν να κινούνται οι άνθρωποι στην κοινωνία και στο χώρο. Γι' αυτό πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα μέτρα για αυτό. Δεύτερον, κάτι το οποίο είναι σημαντικό σε αυτά τα οποία είπατε, υπάρχει μια διαρθρωτική ανεργία, έλλειψη ανθρώπων που θα, είναι, θα έχουν τα προσόντα για αυτά τα 7 εκατομμύρια θέσεις που είπατε κυρία Ροντρίκε. αλλά έχετε και εσείς κυρία Φούξ δίκιο, υπάρχουν γυναίκες με προσόντα αλλά δεν έχουν τις ευκαιρίες. Εκεί πέρα λοιπόν πρέπει να δουλέψουμε για να ανοίξει να ανοίξουν κάπως ε, αυτοί οι διάδρομοι γιατί 54% των πτυχιούχων είναι γυναίκες αλλά μετά σε επιχειρήσεις που είναι, εξαφανίζονται. Γιατί πρέπει να βρούμε μια απάντηση. Μετά ένα άλλο ερώτημα το οποίο δεν με απασχολεί και δεν έχω κάποια απάντηση και ελπίζω να λάβω. Κύριε Ροντρίγκης, ε, κύριος, Πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας για τους ανθρώπους, δεν επιτρέπεται να είναι πολύ ακριβές ταυτόχρονα όμως μπορούμε να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στις υπηρεσίες για ηλικιωμένους ανθρώπους ε, στον τουρισμό, στον πολιτισμό ε, θέσεις όμως οι οποίες κοστίζουν απ' την άλλη γιατί σημαίνουν πολλά προσόντα και έχουμε άρα δύο αντιφατικές ε, τάσεις. Τα τελευταία 20-30 χρόνια δηλαδή στην οικονομία πηγαίναμε προς την κατεύθυνση του ότι όσο περισσότερη οικονομική δύναμη ε, είχε μία επιχείρηση, τόσο περισσότερους ανθρώπους απέλυε για να τους αντικαταστήσει με μηχανές ή για να γλιτώσει κόστος. Εδώ πέρα έχουμε μία αντίφαση λοιπόν ε, και η οποία πρέπει να απαντηθεί και πρέπει να απαντηθεί ε, ε, συγγνώμη, δεν έχουμε συχνά τόσο πολλούς ομιλητές για να δούμε πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτά τα πράγματα. Θυμάμαι κάτι που λέγαμε στη Γερμανία πριν από 30 χρόνια. Πέρα από τον φόρο κύκλου εργασίων ή π.χ τον φόρο στις ε, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, μπορούμε να βάλουμε ένα φόρο μηχανών, λέγαν τότε. Δεν ξέρω, σκέφτεσαι κάτι τέτοιο. Κυρία Χολμάια, κύριε Πρόεδρε, με εκπλήσει το ότι μιλάμε ακόμα για... και μπερδεύουμε τα εμπορικά ισοζύγια με τα ισοζύγια πληρωμών. Ε, σε μια τέτοια εποχή δηλαδή το εμπορικό ισοζύγιο δεν είναι, χωρίς να θέλω να απευθύνω κάποια κατηγορία προς την Ολλανδία, δεν είναι δυνατόν αυτό το πράγμα ε, να λέμε ότι είναι κακό το ότι έχει καλό εμπορικό ισοζύγιο η Ολλανδία, το καλύτερο στην Ευρώπη. Πρέπει να δούμε γενικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι θα κάνουμε, βέβαια, ποιον θα βοηθήσουμε, να βελτιώσουμε την κατάσταση. Ε, και όχι να κάνουμε αυτό το οποίο συνηθίζουμε στην Ευρώπη, να ασκούμε κριτική στου καλύτερου την Ολλανδία δηλαδή εδώ πέρα και να δούμε πώς θα φέρουμε αυτούς προς τα κάτω. Ε, δεν μας βοηθάει αυτό. Το ερώτημά μου τέλος πάντων πάει σε μια άλλη κατεύθυνση. Άκουσα αυτά τα οποία είπατε για την εμπιστοσύνη και πράγματι οι ΙΠΑ έχουν φοβερή αυτοπεποίθηση. Εμείς έχουμε συνέχεια αμφιβολίες στην Ευρώπη. Οι Αμερικανοί στη χειρότερη κατάσταση έχουν την βεβαιότητα πώς θα τα καταφέρουμε, μπορούμε, μόνοι μας θα βγούμε από τις δυσκολίες και τα λοιπά. Δεν υφίσταται σε μας κάτι τέτοιο. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι πρώτον, μήπως δεν χρειάζεται, μήπως χρειάζεται στον τομέα της παραγωγής να προσπαθήσουμε εντός της Ευρώπης να επενδύσουμε όχι μόνο στην πράσινη τεχνολογία αλλά και στην πράσινη τεχνολογία. Στις σύγχρονες τεχνολογίες γενικά που έχουμε διάφορα ισχυρά σημεία στην Ευρώπη. Η ιατρική τεχνολογία, η βιοτεχνολογία, κάθε χώρα έχει το ισχυρό της σημείο. Να τα συνδέσουμε αυτά στην εσωτερική αγορά αντί να φεύγει όλη η παραγωγή εκτός της Ευρώπης και να την εισάγουμε μετά ξανά εμείς. Δηλαδή έχει μετατοπιστεί όλη η παραγωγή στην Ασία. Δεν είναι αυτό α, ισχυρό σημείο της Ευρώπης το να βασιζόμαστε μόνο στις υπηρεσίες. Βλέπουμε το τι σημαίνει αυτό τώρα για την Αγγλία σήμερα. Δεύτερο ερώτημα για εσάς. Όταν μιλάμε για τις δουλειές διαπιστώνουμε πως μιλάμε για παγκοσμιοποιημένες τράπεζες και υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών. Ταυτόχρονα όμως την ίδια ανάσα βλέπουμε πως οι περισσότερες θέσεις εργασίας δημιουργούνται σε μικρομεσαίες και σε μικρές ε, επιχειρήσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Μήπως λοιπόν τονίζουμε συνέχεια και τη φορολογική συζήτηση ε, τα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας ενώ η κοινωνική και η οικονομική σταθερότητα σχετίζεται με τις ε, μικρές επιχειρήσει και έρχομαι στην ερώτησή μου για να μην ανησυχείτε. Μήπω πρέπει να σκεφτούμε ποιες, ποιους φόρους θα έπρεπε να έχουμε αντί να αυξάνουμε τους φόρους για να παρακινήσουμε την οικονομία αντί να λέμε και άλλους φόρους θα επιβάλλουμε στην οικονομία γιατί τελικά όλα αυτά καταλήγουν στους κοινωνικά ασθενέστερους και χάνονται θέσεις εργασίας. Να δούμε δηλαδή πώς θα έχουμε έξυπνους φόρους, όχι μόνο να τους μειώσουμε, αλλά να τους αλλάξουμε κιόλα. Μάλιστα, υπάρχει και για μένα χρόνος. Ευχαριστώ. Θέλω να πω... Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα πάρα πολύ την κυρία Ροντρίγε που τόνισε το πολύ βασικό θέμα της σύγχρονης Ευρώπης που θέλει να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης, αλλά που έχει κατακαιρματίσει τις προσπάθειές της. Ε, ε, χωριστά η καινοτομία, χωριστά η έρευνα, χωριστά η εκπαίδευση. Όλα αυτά όμως πρέπει να συνδυαστούν, γιατί δεν πρέπει να συζητάμε μόνο για καινοτομία και να ξεχνάμε την διαβίου κατάρτιση. Όλα αυτά πρέπει να πάνε μαζί. Αν χρειάζεται καινοτομία, χρειάζεται και κατάρτιση. Έπειτα, εργοδότες, τα συνδικάτα πρέπει μαζί να συνεργαστούν υπέρ της καινοτομίας. Έτσι επιταχύνεται και βελτιώνεται η παραγωγικότητα. Έτσι αλλάζουν οι χώροι εργασίας, οι θέσεις εργασίας, εκεί δηλαδή που δουλεύουν και ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν οι εργαζόμενοι. Πρέπει λοιπόν όντω να είμαστε πιο δημιουργικοί και δεν έχει σημασία, είτε πρόκειται για καθαρίστρια, είτε πρόκειται για έναν μάνατζερ μια μικρή ε, επιχείρηση. Η καινοτομία χρειάζεται παντού και προπόθεση για αυτήν είναι η εκπαίδευση. Έρευνα λοιπόν, καινοτομία, εκπαίδευση πρέπει να τα βάλουμε μαζί. Και εσείς είπατε ότι πρέπει να δούμε τις ε, δημιουργικές επιχειρήσεις. Όντως, ενώ ή για την πληροφορική εμείς δουλεύουμε ή για τη βιομηχανία, γιατί ακόμα βρισκόμαστε στο παρελθόν. Δεν έχουμε αντιληφθεί περί την πρόκειται η νέα οικονομία. Όταν επενδύουμε στις επιχειρήσεις, Επενδύουμε στην αυτοκινητοβιομηχανία, στην ε, χαλιβουργία, σε παλιωμοδίτικες βιομηχανίες. Εγώ μόλις επέστρεψα από τη Νέα Υόρκη. Εκεί ε, μελέτησα λιγάκι τον κλάδο των ε, παιχνιδιών μέσω της πληροφορικής. Είναι μια νέα βιομηχανία που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Οι επενδυτές επενδύουν μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε τέτοια παιχνίδια ηλεκτρονικά. Δεν είναι αποτελεί όμως μέρος της δικιάς μας στρατηγικής εξόδου από την κρίση. Έπειτα, οι υπηρεσίες. Και εκεί μπορούμε να δημιουργήσουμε πολύ περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Πρέπει λοιπόν να αλλάξει η νοοτροπία μας και να απομακρυνθούμε από την ε, βιομηχανία και να πάμε στην κοινωνία της γνώσης. Τέλος για τις γυναίκες. Όταν ε, κοιτάμε την πράσινη οικονομία το 80% είναι οι άντρες και μόνο 20% οι γυναίκες. Λοιπόν θα έπρεπε, όπως λέμε και εμείς στην Επιτροπή Γυναικών, να χρησιμοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτή την κρίση για να πάψει ο κατακερματισμός ανάλογα με το φύλλο στην αγορά εργασίας. Δεν θα μακρηγορήσω για να απαντήσουν και οι ομιλήτριες. Θέλω να επανέλθω σε κάτι άλλο. Καταρχάς την κυρία Ροντρίγκε. Αναφερθήκατε στα απαραίτητα ευρωπαϊκά εργαλεία ε, για τις χρηματαγορές. Τι άλλο όμως. Τι άλλο θα κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να είμαστε σίγουροι ότι αύριο μεθαύριο θα έχουμε μια ανάπτυξη ε, και επενδύσεις που θα δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Στην άλλη ομιλήτρια, η οποία μίλησε για το θέμα της εμπιστοσύνης. Για μένα ένα από τα λάθη που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση στη διαχείριση αυτής της κρίσης και νομίζω ότι είναι η πιο δύσκολη οικονομική έννοια να τη χειριστούμε, είναι το πώς χειρίστηκε το θέμα της εμπιστοσύνης. Ε, ζητώ συγγνώμη για αυτούς που με ξέρουν, γιατί τα λέω συνέχεια αυτά. Το Μάρτιο του 2008 το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για πρώτη φορά λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε ενδεχομένως να μπει σε, σε ύφεση. Εκείνη τη στιγμή στη Γερμανία έχουμε τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2008 που πέφτουν. Μειώνεται Μειώνονται οι πωλήσει στα αυτοκίνητα. Δεν χρειάζεται να είναι κανεί ε, επάγοντα, να καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά. Εγώ τότε ήμουνα υπεύθυνη τη ε, Οικονομική Επιτροπή. Ε, έλαβα ε, ένα τηλεφώνημα τον κύριο Τρισέ, την κυρία Λαγκάρτ, από τον κύριο Γιούνκερ και από τον κύριο Αλμούνια. Αλήθεια σα λέω, ε. Και μου λένε, να τα αμερικανικά στοιχεία του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου που επηρεάζονται από την κατάσταση στην αμερικανική οικονομία. Εμεί μια χαρά τα πάμε. Δεν είναι προσαρμοσμένα στην ευρωπαϊκή πραγματικότητα. Γιατί τα λέγανε αυτά. Γιατί υπήρχε αυτό ο φόβος ότι τα νοικοκυριά θα χάσουν την εμπιστοσύνη και ότι δεν θα καταναλώνουν πια. Επομένως, ομφαλοσκοπούσαμε, ας πούμε, και στρουθοκαμιλίζαμε, ε, κάναμε ότι δεν τρέχει τίποτα. Γι' αυτό ίσως στάσαμε σε αυτή την ε, κρίση σε μορφή W, τη διπλή κρίση. Όντως, αυτό το θέμα της έλλειψης εμπιστοσύνης ε, θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας στρατηγική ανάκαμψης. Και μετά από τη σημερινή ακρόαση, το συμπέρασμα που βγάζω είναι ότι αυτές οι στρατηγικές εξόδου από την κρίση θα πρέπει να είναι πολύ συνετές, πολύ προσεκτικές και θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους διαφορετικά τα διακυβεύματα ε, που συνδέονται με τη μείωση του χρέους. Στο βαθμό που παραμένουμε σε μια δύσκολη περίοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα δύο λόγια για αυτά που υπόθηκαν για την εσωτερική αγορά. Όταν ο Μάριο Μόντι έκανε την πρόταση του, εγώ ήμουνα ενθουσιώδης. Αλλά όσο τον ακούω, ανησυχώ. Γιατί αντίθετα από την κυρία Ροντρίκε, δεν νομίζω ότι το θέμα της φορολογίας είναι το μόνο που θα πρέπει να μας ανησυχεί. Έτσι όπως οικοδομείται η εσωτερική αγορά, ε, το γεγονός ότι δεν υπάρχει εναρμόνιση των φόρων καταστρέφει την εσωτερική αγορά. Και νομίζω ότι η περιοδία στις πρωτεύουσες του κ. Μόντι και τα όσα είπε θα πρέπει να μας ανησυχούν. Για τη διαδικασία της, της Μπολόνιας θέλω να πω κάτι ακόμα. Ε, άλλα πέντε λεφτά σας δίνουν διερμηνείς. Λοιπόν, για τη διαδικασία της Μπολόνιας ε, σπάνια έχουμε την ευκαιρία να, να διαρωτηθούμε για αυτό το θέμα. Στη Γαλλία, ειδικά στον τομέα της έρευνας, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για τη σημασία αυτή της διαδικασίας που έφερε σε αντιπαράθεση τα πανεπιστήμια. Αντί να δημιουργήσει, ας πούμε, δίκτυα ε, αριστείας και εξυπνάδας. Κάτι, κάτι αντίστοιχο με αυτό που υπήρχε το Μεσαίωνα. Τα λέω ελλειπτικά τώρα, αλλά καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Να ζητήσω τις δύο μιλήτριες λακωνικά, όσο πιο λακωνικά μπορούν, να μας απαντήσουν. Γιατί οι διερμηνήσεις θα μας εγκαταλείψουν σε πέντε λεφτά. Ναι. Για τις φορολογικές πολιτικές Έχουμε δύο προβλήματα. Συμφωνώ μαζί σας. Όλοι οι φόροι να πηγαίνουν προς την ίδια κατεύθυνση και από την άλλη να υπάρξει μια σύγκληση, όχι εναρμόνιση, να κλείσουμε την ψαλίδα στο επίπεδο της ε, φορολόγησης. Αυτό είναι το πρόβλημα στην εσωτερική αγορά. Τώρα, τα δημογραφικά προβλήματα. Πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το κίνδυνο που απορρέει από την απώλεια του δημογραφικού δυναμικού θα πρέπει να αυξήσουμε την κινητικότητα και η μετανάστευση είναι και μια λύση για την Μπολόνια. Συμφωνώ ότι μέχρι στιγμής η Μπολόνια βοήθησε να τυποποιηθεί η εκπαίδευση και η παιδεία στην Ευρώπη, αλλά δεν τόνωσε την κινητικότητα. Κάτι λοιπόν δεν πάει καλά. Ήμουνα στην Επιτροπή που ασχολείται της της Ευρωπαϊκής ε, Επιτροπής που ασχολείται με το Εράσμους. Θέλουμε πραγματικές προϋποθέσεις και κίνητρα για να εξαπλωθεί το Εράσμους, να δώσουμε κίνητρα στους φοιτητές κτλ. Τρίτον, έχουμε αυτό το χάσμα από μεταξύ νέων που είναι πτυχιούχοι που έχουν πολλά προσόντα αλλά από την άλλη δεν έχουμε εργάτες που να έχουν αρκετές δεξιότητες. Ε, θα πρέπει να προσαρμόσουμε επίσης και τις δουλειές που δημιουργούνται. Πώς μπορούμε να το κάνουμε. Γι' αυτό θα πρέπει να, να λάβουμε υπόψη μας την καινοτομία και τη διαβίου κατάρτιση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αλλά πίσω από όλα αυτά υπάρχει ένα πρόβλημα εμπιστοσύνη. Συμφωνώ μαζί σας εδώ. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη. Έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα με μια σταθή ανάκαμψη, ο μόνος τρόπος για να δημιουργήσουμε εμπιστοσύνη είναι να υπάρξει μια νέα συμμαχία μεταξύ κράτους και ιδιωτικού τομέα, κρατικής παρέμβασης και ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Το κράτος έχει ευθύνη, πρέπει να δώσει ευκαιρίες με τις κρατικές προμήθειες, με πρότυπα, νέα πρότυπα, με την παροχή οικονομικών μέσων. Από την άλλη χρειαζόμαστε όμως και τον ιδιωτικό τομέα και τις πρωτοβουλίες του. Η κατάσταση είναι τέτοια που δεν μπορούμε να βασιστούμε μόνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Θα πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά. Γι' αυτό χρειαζόμαστε να συντονίσουμε τις πολιτικές που μέχρι στιγμής ήταν ασυντόνιστες. Και είναι απορία άξιων, γιατί δεν συντονίσαμε την βιομηχανική, την εκπαιδευτική πολιτική, την πολιτική έρευνας και καινοτομία. Είναι κατακαιρματισμένες εδώ στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη με ελάχιστε εξαρέσεις. Πρέπει να δημιουργήσουμε λοιπόν ένα άλλο πλαίσιο Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει. Και στην, στα πλαίσια της στρατηγικής της Ευρώπης για το 2020 δεν ρυθμίζεται. Αυτά έτσι πολύ σχηματικά και πολύ ελλειπτικά. Τώρα όμως πρέπει να συνεχίσουμε στα αγγλικά. enough yet about the importance of trust, about how it plays out in the overall economy, and certainly